Dear colleagues, can we start the session? Let's λοιπόν. Just start with saying that the session is web streamed, so... Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται μέσω διαδικτύου, γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε σωστοί, να συμπεριφέρεστε καλά, λέει η Πρόεδρος, και τα λοιπά. Θα ήθελα να καλωσορίσω εκ βάθους καρδίας όλους τους ε, συναδέλφους που έρχονται από τα, Ευρωπα... Ε, συγγνώμη, Εθνικά Κοινοβούλια για να είναι σήμερα μαζί μας. Και θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι σήμερα έχουμε και πρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου που θα μας μιλήσει για πρώτη φορά μετά από την έγκριση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Ε, ο... Έχουμε τον Επιτρόπο Χάν επίσης. Ε, είναι εξαιρετική λοιπόν η ευκαιρία και έχουμε και την ε, κυρία Ιβώνα Βέλντελ η οποία είναι αναπληρωτής υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πολωνία και εκπροσωπεί βεβαίως την Πολωνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε επίσης τρεις συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα μιλήσουν ως κεντρικοί ομιλητές έτσι ώστε να έχουμε ένα έναυσμα, μια κίνηση στη συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Έθνς Κίνσκεν, ο οποίος θα μιλήσει από την Γερμανική Βουλή, τον Bundestag, τον κύριο Λάσλο Χάπης από την ε, Ουγγρική Βουλή και τον κύριο Βίλι Τροφάνικ από την Σλοβενική Βουλή. Θα ήθελα επίσης να δραχθώ της ευκαιρίας έτσι ώστε να εξηγήσω εν συντομία ε, μερικά πράγματα. Θα πούμε και κάποια πράγματα επί της ουσίας. Μετά ο Επίτροπος Ιωάννης Χάν θα πάρει το λόγο, η κυρία Βέντελ και μετά οι τρεις συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μετά βεβαίως θα ξεκινήσει η συζήτηση και θα μπορούν όλοι και μέλη του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να πάρουν το λόγο, να υποβάλουν ερωτήσεις κτλ. Θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να συμπληρώσετε αυτό το έγγραφο έτσι ώστε να ξέρουμε πόσοι θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να το κάνετε επομένω όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να ξέρω πόσους ομιλητές θα έχω εγγεγραμμένο στη λίστα μου. Ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω δύο λόγια. Γιατί δηλαδή αυτή η συνάντηση είναι τόσο σημαντική για μας και είναι τόσο σημαντική για να έχουμε μαζί μας και τον Επίτροπο και την Υπουργό. Κοιτάξτε, η συνεδρίαση αυτή, η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα ιδιάζον και ιδιαίτερο πλαίσιο. Πολλής λόγος γίνεται στην Ευρώπη για ε, σταθερότητα ε, και επομένως θα πρέπει σιγά σιγά να μεταφέρει το βάρος της προσπάθειας ε, και προς την ανάπτυξη γιατί τα <clears throat> επόμενα χρόνια χρειαζόμαστε βεβαίως και παραδοσιακής μορφής ανάπτυξης αλλά και νέους φορείς ανάπτυξης. Θέλουμε επενδύσεις και οι επενδύσεις όπως όλοι γνωρίζουν χρειάζονται χρηματοδότηση και επομένως η εξέβρεση των χρημάτων, των κονδυλίων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κατά αυτή την έννοια, ο μελλοντικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιετές πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών για την επόμενη επταετία, βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σκέλος της δημόσιας χρηματοδότησης. Έχουμε ακόμα δύο χρόνια που υπολείπονται και σε αυτά τα δύο χρόνια θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο προϋπολογισμός θα είναι τέτοιος ώστε να μπορέσει να ελκύσει ιδιωτικό χρήμα. Θα πρέπει να επενδύσουμε επίσης τα, τις ευρωπαϊκές πιστώσεις, τα ευρωπαϊκά κονδύλια μάλλον, σε ε, νέες επενδύσεις ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά επενδύσεις οι οποίες θα ακολουθούν ένα διαφορετικό καινοτόμο ε, σχήμα ε, και που θα οδηγήσουν σε σταθερές δουλειές, ε, που θα οδηγήσουν σε αναστροφή της τάσης απώλειας των θέσεων εργασίας κτλ. Με την απόφαση της Επιτροπής ε, όσον αφορά την έγκριση της νέας δέσμης της νέας πολιτικής είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ μαζί μας τον Επίτροπο κύριο Χάν να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι περιέχει αυτή η νέα δέσμη και επίσης να δούμε παράλληλα και πώς εμφανίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Το, κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μάλλον περιορισμένο ρόλο ε, ε, στον πολιετή προγραμματισμό ε, αλλά βεβαίως μπορεί να ακουστεί η φωνή μας πάρα πολύ δυνατά όσον αφορά τον μελλοντικό προϋπολογισμό και αυτό θα κάνουμε. Και άλλωστε είναι και ο νέος ρόλος, ο διευρυμένος που έχει το Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και υπάρχει, μην ξεχνάτε, και αυτή η διαδικασία συναπόφασης, η co-decision, ε, όπου ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντικός και αναβαθμισμένος σε σχέση και με το Συμβούλιο. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Έχουμε δουλέψει με τους ε, συνεργάτες του Επιτρόπου κυρίου Χάν. Τα τελευταία δύο χρόνια δουλέψαμε πολύ με τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο που ασχολείται δηλαδή με την ε, περιφερειακή ανάπτυξη, έχουμε μάθει ε, να γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, ε, να υπάρχει πλέον ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και έχουμε δουλέψει πολύ μαζί. Επίσης να πω ότι σε συνεργασία με το Συμβούλιο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει την εργασία του για την, ε, με την ε, Τρόικα. Επομένως δεν δουλεύουμε μόνο με την Πολωνική Προεδρία, αλλά και με, την, με τις μελλοντικές προεδρεύουσες χώρες Δανία και Κύπρο έτσι ώστε να καθορίσουμε ένα στέρεο πλαίσιο συνεργασίας. Και εδώ έρχεστε εσείς, ο δικός σας ρόλος. Θα ήθελα επομένως να επιβεβαιώσω ότι για αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο έχετε την, πράσινη, έχετε την ε, ε, κίτρινη κάρτα στο χέρι σας, αλλά θα πρέπει να την χρησιμοποιήσετε με σοφία και σύνεση λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομίες των χωρών σας και την ευρωπαϊκή οικονομία. Βεβαίως είμαστε όλοι εδώ στη διάθεσή σας έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να εξηγήσουμε κάτι που δεν έχετε ενδεχομένως καταλάβει και βεβαίως να στηρίξουμε αυτήν την περιφερειακή πολιτική η οποία θα δημιουργήσει, θα γεννήσει ανάπτυξη. Αυτά ήθελα να σας πω και να ζητήσω επομένως από τον Επίτροπο κύριο Χάν να μας πει δύο λόγια ή λίγο παραπάνω από δύο λόγια ε, για το νέο πλαίσιο. Ε, κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ντανούτα, ευχαριστώ πολύ καθηγητή, κυρία Χέμπνερ, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως θα ήθελα να καλωσορίσω, μια και ακούγεται η συνεδρίασή μας μέσω διαδικτύου, να καλωσορίσω λέγω όλους τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι πράγματι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε διάφορους ε, κανονισμούς που αφορούν τα διορθωτικά ταμεία και που έχω την ευκαιρία λοιπόν να κάνω μια πρώτη παρουσίαση αυτών των νομοθετικών προτάσεών μας για μια νέα πολιτική συνοχής ενώπιον αυτής της ε, ε, διακοινοβουλευτικής επιτροπής. Η Ευρώπη ε, έχει οικοδομηθεί για όλους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Τανούτα Χίμπνερ ειδικότερα. Ανοίγουμε σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική συνοχής. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο το ανέφερε άλλωστε. Οι σημερινές προτάσεις ε, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανανεωμένης Ευρώπης. Ε, νέα, σύγχρονη πολιτική επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο επιγόντως χρειάζονται οι οικονομίες μας, οι πολίτες μας, αλλά και το περιβάλλον μας. Αυτή η σύγχρονη επενδυτική στρατηγική ε, δεν αφορά μόνο εμένα, δεν το σκέφτομαι εγώ δηλαδή μονάχα τις νύχτες που ίσως δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά όλοι μαζί μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία αναφέρθηκε και η Ντανούτα, με πολλές επαφές ε, τυπικές, άτυπες, επίσημες, ανεπίσημες, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ειδικά όμως αυτή η Επιτροπή και ορισμένοι από τους παριστάμενους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων τα μάλα έχουν στηρίξει τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό λοιπόν δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω ενθέρμως όλους. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να πούμε ότι ξεπληρώνονται, έχουν αντίκρισμα οι προσπάθειές μας. Ε, βεβαίως ε, αυτό ισχύει για μένα γιατί η δικιά σας αποστολή μόλις τώρα ξεκινάει όπως είπε και η Ντανούτα. Τώρα ξεκινούν ε, οι μεγάλες ευρείες διαπραγματεύσεις όμως Νομίζω ότι το σημερινό επίτευγμα αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει όλοι από κοινού τον τελευταίο χρόνο. Θυμάμαι ότι πολλοί μεταξύ ημών με υψηλών ε, είχαν δυσκολίες στην αρχή ε, αλλά η πολιτική συνοχή ε, βεβαίως ε, στέφεται τελικά από επιτυχία. Έχουμε 84 περιοχές σύγκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά στοιχεία. Ενώ στο μέλλον θα έχουμε μονάχα 68 περιφέρειες σύγκλησης. 34 εκατομμύρια δηλαδή πολίτες της Ευρώπης είναι τώρα σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει όπως αναφέρονται και όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα του, ε, του πέμπτου πλαισίου, εμείς ε, έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να έχει μια πολιτική συνοχή η οποία θα οδηγήσει στην στρατηγική της Ευρώπης 2020 και βεβαίως θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και σε νέες θέσεις Παρόλα αυτά και παρά τις προόδους που έχουν έχουν σημειωθεί. Βεβαίως η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο. 36 δις ε, δηλαδή ε, περισσότερα χρήματα από την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί σε υποειλοποίηση προγράμματα. Βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ακόμα μερικά πολύ σημαντικά βήματα που μας περιμένουν μέχρι την τελική έγκριση. Βεβαίως ε, δεν αρχίσαμε, όπως είπε και η Ντανούτα, δεν ξεκίνησαμε από το μηδέν. Η ίδια η Ντανούτα ως παλαιά επίτροπος είχε ε, πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις ε, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας και πολλές από αυτές είχαν επιτυχή, ευτυχή έκβαση. Είναι σαφές βεβαίω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα, κυρίω ε, σε, σε αυτά τα χρόνια, σε αυτούς του καιρού ε, ε, του δημοσιονομικού περιορισμού. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα, επομένω καλύτερη συγκέντρωση, καλή εφαρμογή του συστήματος ερεσιμότητας, καθώς επίσης και σωστή κινητροδότηση. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ο, ο χώρος και η δυνατότητα ε, ε, επιλογών ε, που είναι απαραίτητη για ειδικέ περιφέρειες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά δημογραφικά ή γεωγραφικά. Καλύπτουμε βεβαίως κάθε είδους περιφέρεια, αλλά το κύριο μέλημά μας είναι οι πιο φτωχές περιφέρειες. Ε, ε, εμείς δώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερα. Τους βοηθούμε να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους έτσι ώστε ως ο ασθενέστερος κρίκος της Ευρώπης να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της αντοχής ε, ολόκληρης της Ευρώπης και βάσει της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς γνωρίζομαι ότι ένα ευρώ το οποίο ε, δαπανάται στην Πολωνία ε, επιστρέφει 46 cents ε, στην Ευρώπη των 15. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε καλά ότι οποιαδήποτε πολιτική μας έχει οπωσδήποτε μεγάλο αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί ως προς την απλούστευση των κανόνων. Ε, γίνεται μια προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης του συνολικού πλαισίου. Προτείνουμε λοιπόν εναρμόνιση ε, των κανόνων, όχι μεταξύ των διαφόρων σκελών των ιδιωτικών ταμείων, αλλά και όσον αφορά την συνέργεια με την πολιτική ανάπτυξη, σε την πολιτική γεωργίας και θαλασσίων πόρων. το ε, πέντε ταμεία ε, είναι αυτά τα οποία πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ των οποίων ε, το Ταμείο της Γεωργικής Ανάπτυξης, το Ταμείο για την Αλληλεία, το Κοινωνικό Ταμείο κτλ. Αυτή η συνέργεια των πέντε ταμείων θα οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό και για πρώτη φορά καταφέρνουμε να καλύψουμε αυτή αυτά τα ε, ε, ταμεία και να έχουν λοιπόν αυτά τα, τα πέντε ταμεία μια κοινή διακυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, ε, μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων έτσι ώστε η εποπτεία και το σύστημα αναφοράς όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας να είναι πιο σαφές. Θα δείτε αργότερα και πολλές, πολλά παραδείγματα. Δεν θέλω τώρα να βαρύνω την συζήτηση παρά την ε, ε, παρούσα δυσχερή οικονομική κατάσταση ε, έχει καταστεί σαφές και φαίνεται και στο πρόγραμμά μας ότι χρειαζόμαστε καλή επενδυτική περιφερειακή πολιτική έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανάπτυξη, να βελτιώσουμε την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εν τέλει όλες οι περιφέρειες ανεξάρτητα από το βαθμό ανάπτυξής τους θα πρέπει να εστιάσουν την ε, ε, προσοχή τους ε, για να επιτύχουν ολοκληρωμένη έξυπνη ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, να ε, σταματήσει η ανάπτυξη είτε στην συγκεκριμένη περιφέρεια η ανεργία είναι του 8% ε, είτε είναι 20%. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τους πολίτες της Ευρώπης. Φυσικά, σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας δώσω λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία για κάθε περιφέρεια. Αυτό θα γίνει αφού ε, ε, θα έχουμε την τελική συμφωνία για τον προϋπολογισμό των επόμενων ε, των επόμενων προοπτικών. Έχουμε όμως κάποιες προσωμιώσεις. Κυρίως ε, πρέπει να σημειώσω τώρα ότι μέσω των ε, μεταβατικών ε, περιοχών, περιφερειών έχουμε πλέον μια καλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο. Πού πάνε τα χρήματα η συνθήκη αναφέρει σαφώς ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια έτσι ώστε να μικρύνουν ε, οι αποστάσεις ε, ε, μεταξύ των και οι διαφορές μεταξύ των περιοχών και των περιφερειών. Εγώ θέλω η πολιτική συνοχή να γίνει ένα εργαλείο σημαντικό για την Ευρώπη 2020 αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα βασίζεται σε λίγε μόνο πρωτοβουλίε, οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τη την στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, ε, έχοντας κατά νου την Ευρώπη 2020 αλλά δίνοντας στις περιφέρειες την απαραίτητη ευελιξία την οποία χρειάζονται έτσι ώστε να εργαστούν βάσει των ειδικών αναγκών τους. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 35% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 40% ε, στις μεταβατικές και 52 σαν αναπτυγμένες. Ε, νομίζω ότι ε, είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μικρό αριθμό ε, προτεραιοτήτων που οπωσδήποτε θα περιλαμβάνουν την εδαφική χωρική συνεργασία ε, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο εμείς οργανώνουμε τη μελλοντική χρηματοδότηση. Προτείνουμε κοινό στρατηγικό πλαίσιο για πέντε ταμεία που ε, μεταφέρει ακριβώς ε, τους ε, στόχους και τις κατευθύντες γραμμές για την Ευρώπη 2020. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό, να δώσουμε όμως στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν πολυτομιακά προγράμματα τα οποία θα αφορούν πολλά ταμεία όσον αφορά το στρατηγικό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη μέσω λειτουργικών προγραμμάτων θα προχωρήσουν ε, σε διακρατικές ε, συνεργασίες. Βεβαίως προβλέπονται και διαφορετικά ε, επίπεδα διακυβέρνησης, κυρίως σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό. Γι' αυτό ακριβώς ε, προγραμματίζουμε τον, ε, την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών όσον αφορά την, την διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων και τις διαπεριφερειακές συνεργασίες. Ε, υπάρχει και το σχετικό εγχειρίδιο το οποίο αναφέρει το φάσμα και ε, το πλαίσιο εφαρμογής του κάθε ε, ταμείου ας πούμε προγράμματα τα οποία αφορούν την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι τη δημιουργία νέων business models. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ε, σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη ε, και βεβαίως μπορούμε αργότερα να εξειδικεύσουμε τα μέτρα αναφερόμενοι στα μεμονωμένα ταμεία. Όλα αυτά όμως δεν είναι αρκετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ίδια τα κράτη-μέλη, οι ίδιες οι περιφέρειες στην αρχή της προγραμματικής περίοδου ε, να ε, ε, υποβάλουν σαφείς και σαφώς μετρήσιμους στόχους έτσι και να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πρόοδο υλοποίησης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Επίσης, η καλή επίδοση ε, σχετίζεται και με τις σωστές ε, προϋποθέσεις και τους σωστούς όρους. Ε, η αιρεσιμότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να δούμε εάν οι συνθήκες υλοποίησης και δαπάνησης των πόρων είναι σωστές. Προτείνονται λοιπόν κάποιες συμμετρικές γενικές ε, προϋποθέσεις ε, που θα πρέπει να ελέγχονται πριν από την αρχή έναρξη υλοποίηση οποιοδήποτε προγράμματος. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται ρητά και σαφώς έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγάλη διαφάνεια και να μπορεί να γίνει και ο εκ των υστέρων έλεγχος. Μπορώ ας πούμε εδώ να αναφέρω την ε, ε, ύπαρξη στρατηγικών έρευνας ε, που υπάρχουν ήδη σε, που υπάρχει ήδη επίσης το νομικό πλαίσιο για τις μικρές επιχειρήσεις Small Business Act Επίσης, ε, ε, η δυνατότητα ε, κοινή τιμολογιακής πολιτικής για το νερό. Διάφορες αρχές που θα διέπουν την αγορά εργασίας κλπ. Όσον αφορά την αιρεσιμότητα εξπόστ, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα επιβράβευσης ε, των προγραμμάτων που έχουν πάει καλά. Εδώ δεν θέλουμε να εντείνουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των προγραμμάτων. Απλώς θέλουμε προγράμματα τα οποία θα ε, επιτύχουν τον σωστό στόχους ε, και βεβαίως επιβραβεύεται ε, η καλή ε, επίδοση. 5% των πόρων θα δοθούν το 2019 στα προγράμματα τα οποία έχουν λειτουργήσει καλά και εδώ βεβαίως θα ήθελα να ζητήσω εν θέρμος την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζοντας ότι αυτή δεν είναι μια ιδέα που σημερίζονται ε, Γενικώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, προτείνουμε να δημιουργηθεί ισχυρός δεσμός ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και την γενικότερη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής δυσχέρειας ε, ε, η πολιτική συνοχή και τα κονδύλια που σε αυτήν, ε, με αυτήν συνδέονται να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει επίσης ε, να, να ε, σταματήσει ε, η εκροή κονδυλίων τα οποία δεν έχουν αποτελεσματική χρήση ή η χρήση τους δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Βεβαίως αυτό θα είναι ένα, τελική, ένα μέτρο στο οποίο θα προσφύγουμε σαν ε, τελικό μέτρο. Ε, το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των ε, φορέων. Αυτά θα τα δείτε βεβαίως αναλύοντας το έγγραφο το οποίο σας έχει υποβληθεί. Θα πω δύο λόγια τώρα για τα ταμεία για τα οποία είμαι υπεύθυνος. Η βασική ιδέα είναι να προωθεί η ανάπτυξη και η διαθεωρητική προσαρμογή των καθυστερημένων περιοχών. Θα πρέπει να συμβάλλουν στην, στην των στόχων της, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Βασική είναι η ενίσχυση της εδαφικής ε, περιφερειακής συνοχής η υποστήριξη επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό προς επίτευξη στόχων. Καταρχήν σε καθορισμένους ε, σκοπούς επένδυση. Υπάρχουν τρεις συμμετρικές προτεραιότητες που είναι υποχρεωτικές. Καινοτομία, έρευνα, ε, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεταμόρφωση προς μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Ε, τα κονδύλια θα πρέπει να επενδυθούν λοιπόν σε αυτούς τους τρεις ε, στόχους όπου τουλάχιστον 20% των κονδυλίων θα πρέπει να χωρηθούν για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφερειακές ε, περιοχές θα πρέπει 6% να δοθούν για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας ε, λόγω ακριβώς των ε, διαφορών μεταξύ των περιοχών. Το Ταμείο συνεχίζει, θα συνεχίσει να υποστηρίζει προγράμματα σε όλες τις ε, χώρες. Επενδυτικοί τομείς κλειδί, κλειδιά παραμένουν οι μεταφορές. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα νέα εργαλεία. 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια από τα 27 θα πρέπει να δοθούν σε αυτό το νέο μέσο. Η εδαφική συνεργασία, κάτι το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την Επιτροπή και γι' αυτό ακούσαμε πολλές φωνές να καλούν για αύξηση της εδαφικής συνοχής και της εδαφικής συνεργασίας. Γι' αυτό ε, προτείνουμε μία αύξηση της τάξης του 30%. Επίσης, και αυτό θα συμβάλλει σε μία γενική όφηση για επένδυση δημιουργία και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εφαρμογή των συμμετρικών αρχών ανάπτυξης. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίες, αλλά αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να απευθύνονται σε πολύ ε, συγκεκριμένα θέματα. Ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προσθέσουμε εκεί όπου μπορούμε. Για παράδειγμα, τώρα προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ένα ε, ενίο σετ κανόνων ανεξάρτητα από το πού λαμβάνουν χώρα οι δαπάνες. Επίσης ε, προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τις δομές ε, της διαχείρισης, ούτε, ούτε ώστε τα ευρωπαϊκά προγράμματα να έχουν μία ενία αρχή διαχείρισης και μία ενία αρχή οικονομικού αλέγχου οι πιστοποιημένες αρχές ε, δεν θα υπάρχουν πλέον. Ως προβλέπεται στον κανονισμό, αυτό το χρόνο ε, υπήρξε μία αναθεώρηση της ε, πολιτικής και η αναθεώρηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνέχεια είναι ιδιαίτερα σημαντική και Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστούν κανόνες, κάποιοι κανόνες και η πρότασή μας είναι να δοθούν στις χώρες μέλη έξι μήνες ούτε ώστε να βελτιώσουν τις πολιτικές τους. Ταυτόχρονα έχουμε θεσπίσει ένα περαιτέρω στοιχείο ευελιξίας διευρύνοντας το φάσμα ε, δράσης. Πλούστευση. Πολλοί ρώτησαν ε, κατά πόσο μπορούν οι παλαιοί κανόνες να πλουστευθούν. Εγώ θα προτείνω κάποια συγκεκριμένα μέτρα πλούστευσης στο πλαίσιο του νέου προπολογισμού και ιδιαίτερω στο νέο ε, πακέτο. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην εναρμόνιση των κανόνων επιλεξιμότητας, ε, θέμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω. Επίση υπάρχει διεύρυνση τη χρήση του ψευμένου κόστου. Επίση, θεσπίσαμε ε, την ε, δυνατότητα στα, για τα προγράμματα να υποβάλλονται κάποια έγγραφα κάθε χρόνο, ε, μειώνοντας ε, τον τεράστιο διοικητικό άχθος. Επίσης, διευρύνουμε τη χρήση τεχνολογιών ε, πληροφορικής όσον αφορά την συνολική διαχείριση, ούτως ώστε να εφαρμοστεί μια συνεκτική πολιτική. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεγγύης, ούτω ώστε να ολοκληρώσουμε το πακέτο μας, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το ε, Ταμείο Ελεγγύης. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στο Συμβούλιο, κάποιες δυσκολίες στο πλαίσιο του προπολογισμού σε πολλές χώρες μέλη. Γι' αυτό εγκαταλείψαμε την ιδέα να αναζωογονήσουμε την πρόταση του 2005 και καταλήξαμε σε μια νέα πρόταση, η οποία αντανακλά καλύτερα τις παρούσες προϋποθέσεις. Προτείναμε να περιοριστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης μόνο στις, να περιοριστεί στις φυσικές καταστροφές, περιλαμβάνοντας όμως ε, τις ε, επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στον χώρο της υγείας ε, και που προωθούν από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Και επιπρόσθετα καλύπτει περιπτώσεις ξηρασίας. Ε, επίσης υπάρχουν και άλλα σημαντικά κριτήρια για τις φυσικές καταστροφές που βασίζονται στο ε, ποσοστό του, ε, ε, στο ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας. Και καταβάλλεται η προσπάθεια να εκπληρωθούν τα κριτήρια σε συνάρτηση με τη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης θα επιταχυθούν κάποιες πληρωμές, ε, θεσπίζοντας τις ε, πληρωμές προκαταβολών ενώ θα περιορίζονται οι χορηγίες σε απόλυτους όρους. Επίσης θέλουμε οι χώρες μέλη να προσπαθήσουν να θεσπίσουν κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις ε, που να τις συνδέσουν με τις πληρωμές σύμφωνα με την, ε, σε συνάντηση πάντοτε με την εφαρμογή της σημαντικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Η, προπαρασκευή των, η πρόληψη των φυσικών καταστροφών ε, θα πρέπει να συνδεθεί με την ε, εκταμείευση των κονδυλίων για την αποτροπή των καταστροφών ή την επανόρθωση των καταστροφών. Και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο όλων αυτών μπορούν να σημειωθούν σημαντικές πρόοδοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σας έδωσα μία ματιά, μία εποπτεία της συνολικής πολιτικής συνοχής και τώρα εναπόκειται σε εσά τους ε, εκπροσώπους ε, των περιφερειών, ούτω ώστε να συμβάλλετε επικοδομητικά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τους προσεχείς ε, μήνες. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την ανταλλαγή απόψεων ε, στο πλαίσιο της συζήτησης και θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω τυχόν ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Ε, Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ε, όλοι μας ε, περιμέναμε ε, το νομοθετικό πακέτο για την Ευρώπη 2020 Πολλοί αναμένουμε ανυπομονησία να δουν τις λεπτομέρειες μιας από τις πιο σημαντικές μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπη σκιαγράφησε στην, την ανακοίνωσή της για τον προϋπολογισμό τον Ιούνιο αυτού του έτους. Παρόλο που όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ βραχυπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε την πολιτική συνοχής από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να εργαστεί με πολύ γρήγορο ρυθμό. Αυτό θα ήθελα να το πω ευθύ εξ αρχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει προθυμία συνεργασία εκ μέρου όλων των εταίρων μα. Εκ μέρου τη Πολωνική Προεδρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Χάν για την παρουσίαση των νέων ε, στόχων της πολιτικής συνοχής και έχουμε επίγνωση ε, πόσο νομοθετικό άθος προποθέτει αυτή η προσπάθεια της Κομισιόν. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας ε, συζήτησης, έντονης συζήτησης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και γνωρίζουμε τι είδους δυναμισμό είχε αυτή η συζήτηση, αυτή η αντιπαράθεση και πόσες διαφορές υπήρξαν μεταξύ των προσεγγίσεων των διαφόρων χωρών μελών. Ε, το μέλημα αυτό δυσχεράθηκε ακόμα περισσότερο από την παρούσα οικονομική συγκυρία και την οικονομική κρίση, τι οποίε, τις επιπτώσεις, οι επιπτώσει είναι ακόμα αισθητέ. Θεωρούμε ότι οι προτάσει ε, τη Επιτροπής είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τη διαδικασία διαπραγμάτευση. και ελπίζουμε ότι θα είναι σύντομε οι διαπραγματεύσει και θα καταλήξουν σε έναν ικανοποιητικό για όλε τι πλευρέ συμβιβασμό. Οι προτάσει μοιάζουν να είναι ισορροπημένε και να αντανακλούν τα σημαντικότερα θέματα τα οποία τέθηκαν στις διάφορες συζητήσεις. Αυτό το οποίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι το κοινό όραμα της πολιτικής συνοχής, μια σύγχρονης πολιτικής, η οποία θέλει να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της ε, σύγχρονης ε, εξέλιξης και θέλει να είναι μια, αποσκοπημένη είναι μια πολιτική κοντά στον πολίτη. Κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργολείο κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 και άλλωστε από αυτό το πρίσμα παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι εισακούστηκε η φωνή των χωρών μελών υπό την έννοια μιας προσέγγισης που βασίζεται περισσότερο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενώ και η πολιτική αυτή είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η προγραμματική στρατηγική με το στόχο να συνδεθεί η πολιτική συνοχής με την οικονομική πολιτική. Μία βιώσιμη περιφερειακή πολιτική μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εφόσον ε, κάποια τομεακά διαφορετικά μέτρα ε, συνενωθούν σε μια ενιαία στρατηγική. Με τον τρόπο αυτό συμπληρωματικά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν μια ενιαία δέσμη και μπορούν να απομακρυνθούν τα αντιφατικά μεταξύ τους μέτρα. Μια ε, προσέγγιση της πολιτικής η οποία να αποσκοπεί σε αυτά αποτελέσματα θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διατύπωση συγκεκριμένων όρων και θα πρέπει να είναι συντονισμένη όσον αφορά το περιεχόμενό της. Θα πρέπει οι χώρες μέλη να έχουν τη συνέντευξη ότι η επίτευξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων δεν συνιστά ε, κύρωση, αλλά είναι η ε, προσπάθεια Αύξηση τη ε, αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων συνοχής. Και στο πλαίσιο αυτό παραμένει σημαντικό να εξασφαλιστεί η ευελιξία στο επίπεδο του προγραμματισμού για τις διάφορες χώρες. Έχουμε την πεποίθηση ότι η πρόταση της Επιτροπής πρόκειται να ικανοποιήσει αυτές τις προσδοκίες. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το γεγονός ότι έχουν προταθεί διάφορες ενδιαφέρουσες ε, λύσεις οι οποίες ε, συμφωνούν με την ε, εδαφική αλλά και την αστική, την περιφερειακή αλλά και την αστική διάσταση. Και αυτό, αυτή είναι πολύ σημαντική η πτυχή της προσέγγισης αυτής. Ε, μεταξύ των χωρών μολών έλαβε χώρα μια πρώτη ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων υπό το πρίσμα των ανακοινώσεων της Επιτροπής τον Ιούνιο και μας επισημαίνει ότι ορισμένα θέματα απαιτούν μια περαιτέρω βάθος ανάλυση. Από τις ε, διάφορες συζητήσεις σε σχέση με την εξυγίανση προκύπτει ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί το Connecting Europe ε, Facility με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνεχής. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ε, κατηγορία υποστήριξης για ορισμένες ε, αποκλεισμένες περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μακροοικονομική διαχείριση, ειδικά ανακύπτει το ερώτημα πώς η Πολωνική ε, Προεδρία θέλει να διαμορφώσει τις διαπραγματεύσεις. Εκ παραδόσεως, οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται στο επίπεδο των ομάδων εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον αφορά τα διορθωτικά κονδύλια. Ε, στις 12 και στις 13 ε, Οκτωβρίου στις διαβουλεύσεις θα συνεδριάσουν οι ομάδες εργασίες και στη συνέχεια ε, θα παρουσιαστεί το πακέτο των μέτρων από τον κύριο Χάν. Μετά την ολοκλήρωση του γύρου διαπραγματεύσεων και αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποβάλλει στις ε, χώρες τις προτάσεις της, η Πολωνική Προεδρία θα αναφερθεί άμεσα, θα περάσει άμεσα μάλλον στις ε, διαπραγματεύσεις, ούτω ώστε να μπορούμε να ε, αναμένουμε οι χώρες μέλη να κάνουν μια ε, ανάλυση και να τοποθετηθούν. ήδη έχει Ήδη θέλουμε να επιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία και οργανώσαμε ένα σεμινάριο με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 14 Οκτωβρίου με θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό. Εν ώψη των ε, διακοπών της Πάψης των Χριστουγέννων ε, θα υπάρξει μια στενότητα χρόνου γιατί μας μένουν μόνο δύο μήνες. Άρα λοιπόν ε, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εντατικό γύρο 11 συνομιλιών που θα αφορούν τα θέματα της διατύπωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, της περιφερειακής ανάπτυξης και άλλα προβλήματα περιφερειακής συνεργασίας. Ο στόχος μας θα είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, ώστε η ιδανική και η Κυπριακή Προεδρία να μπορέσουν να εστιάσουν τη δική τους προσοχή σε άλλα θέματα έχουμε την ε, πρόθεση μέσω μιας έκθεσης της Πολωνικής Προεδρίας να αναφερθούμε στα σημαντικότερα στρατηγικά θέματα τα οποία στη συνέχεια θα ε, τεθούν υποσυζήτηση στους αρμόδιους ε, υπουργούς σε μια επίσημη συνάντηση στις 16 12 και ελπίζουμε ότι η ανάλυση μιας δέσμευσης των ε, ηθινόντων θα προσδώσει σε όλη τη διαδικασία αυτή μια δυναμική διάσταση. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ε, ε, ήδη θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει σε, διάφορες, σε διαφόρους γύρους συνομιλιών και σε διάφορες ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων με, με εσάς έχουμε δείξει ότι για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός εταίρος, είναι και παραμένει. Γι' αυτό πάντοτε τίνουμε δίκον ου στην φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε την πρόθεση τακτά χρονικά διαστήματα να συναντιόμαστε με τους εισηγητές και τις ηγήτρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και να τους προσκαλούμε στα δικά μας σεμινάρια για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είμαστε επίσης στεναρά πεπισμένοι ότι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών θα επιταχύνει την ψήφιση αυτού του κανονισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα um, ήθελα Θέλω να καλέσω τον εκπρόσωπο του Bundestag να πάρει το λόγο της Γερμανικής ε, Βουλής. Αγαπητέ ε, κύριε, αξιότιμα κύριε Χάν, αγαπητοί συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί θα θέσουμε το πλαίσιο για τα έτη από το 2014 στο 2020 και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των μελών τη και έχει τώρα 27 μέλη. Δεν είναι μόνο ο αριθμό των μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξάνεται, αλλά και η ίδια η Ευρώπη εξελίσσεται από κοινού. Και οι ιδιωτικέ συνθήκες στην κάθε χώρα τίνουν προ μια εξομοίωση. Ε, θα ήθελα να σας επισημάνω ακριβώς ε, επειδή ε, έχω μια εμπειρία στην περιφερειακή πολιτική και γνωρίζω πώς ε, άλλαξε η κατάσταση σε διάφορες ε, χώρες. Πριν από 15 χρόνια, για παράδειγμα, σε εμάς στη Γερμανία, οι περιφέρειες, ε, το βαβαρικό δάσος κατά μήκος της, των συνόρων της Τσεχίας ή η οι Άλπις ε, στη Βόρεια Γαλλία, πολύ φτωχές περιοχές με μεγάλο αριθμό ανέργων, ε, πάνω από 14% ανέργους. Και όλα αυτά άλλαξαν ευτυχώς προς το καλύτερο. Και αξιότιμοι ε, συνάδελφοι, ασφαλώς όλοι στις χώρες σας θα γνωρίζετε κάποιες περιοχές, κάποιες περιφέρειες που ε, υπήρξαν στο παρελθόν πολύ φτωχές και τελικά ε, μπόρεσαν να εξελιχθούν και να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις συνθήκες για τους κατοίκους τους. Το γεγονό ότι κάτι τέτοιο επιτεύχθηκε και να ε, κατατείνουν ε, προ μία εναρμόνιση συνθήκε διαβίωση των Ευρωπαίων πολιτών, αυτό είναι ένα συν για τι περιφέρειες, αλλά είναι επίση ένα τεράστιο συν για, το, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο, όσες και επιφυλάξει να έχουν ορισμένοι δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίζουν ότι πάρα πολλές περιοχές μπόρεσαν να υποφεληθούν ιδιαίτερως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να παραγνέσουμε το γεγονός ότι το Ταμείο Συνοχής ε, μεταμόρφωσε πραγματικά πολλές ε, περιοχές που ήταν πολύ φτωχές, ε, ακμάζουσες ζώνες ευημερίες. Κυρίες και κύριοι, χωρίς αμφιβολία, το 2007 μέχρι το 2013 οι περιφέρειες θα κάνουν, κάνουν ένα βήμα προς τα μπρος. Τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στην ε, πολιτική συνοχή ήταν μια πολύ καλή επένδυση στις, ε, ε, όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στην Ευρώπη, αλλά και μια συνεισφορά στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος καθαρός πληρωτής και ο πέμπτος ε, μεγαλύτερος ε, σημαντικός αποδέκτης. Και θα ήθελα να τονίσω και το τελευταίο. Ε, ποιοι είναι οι στόχοι που αποσκοπεί να, να εκπληρώσει η πολιτική αυτή. Κατά την άποψή μου είναι τρεις αυτοί οι σκοποί. Πρώτον η σύγκληση για περιοχές που έχουν λιγότερο από το 70% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να προθεθούν και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Γι' αυτό εδώ ε, είναι ιδιαίτερος ε, ισχυρό το αίτημα της πρόθεσης αυτών των περιοχών. Για τις περιφέρειες αυτές που αυτό το κριτήριο, ε, που το κριτήριο μέχρι το 2006 υπάρχει ένα μειούμενο phasing out. Οι υπόλοιπε περιοχές μπορούν ε, να προθεθούν λιγότερο από οικονομική άποψη ε, και να δοθούν ε, χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής για την πρόθεση κυρίως της απασχόλησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας στη Γερμανία για να μειωθεί το χάσμα μεταξύ ισχυρότερων και πιο αδύναμων περιοχών πιο πλούσιων και πιο φτωχών περιοχών. Τρίτον, η εδαφική συνεργασία με τις ε, ε, συνοριακές ε, συνεργασίες θα πρέπει να προωθηθεί στο επίπεδο της περιφερειακής ανάπτυξης. Και θα ήθελα να σε επισημάνω το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μας, ε, έχει πετύχει από μια συνολική άποψη, ολική άποψη. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να οι νέε δομέ ε, ενίσχυση και προώθηση των περιφερειών να προσανατολιστούν στι ήδη φυστάμενε παλαιότερε δομέ. Και οι συνάδελφοί μου στο Γερμανικό Κοινοβούλιο συμμερίζονται αυτή την άποψη. Ε, δύο συνάδελφοι από το Γερμανικό Bundestag, η κυρία Φως και εγώ, και επίσης δύο σημαντικοί πολιτικοί της περιφερειακής πολιτικής, ε, υπουργοί, οι υφυπουργοί από τα κρατήδια, ο κύριος Μάρκοφ και ο κύριος Σνάιντερ, ε, παρίστανται εδώ. Και επειδή θέλουμε να υποβάλουμε τη νέα, ε, επειδή αναμένουμε μάλλον τη νέα πρόταση της Κομισιόν, θα ήθελα να αναφερθώ στα ήδη γνωστοποιηθέντα προγράμματα της Επιτροπής και να πω ότι ήδη Έχουμε ακούσει κάποια πράγματα σήμερα, ε, μέχρι σήμερα από την Επιτροπή. Ε, ε δεν ξέρω αν αυτά θα αποτελέσουν τη βάση αυτού που θα κοινοποιηθεί στις 12 Οκτεβρίου. Ε, 376 δις ε, κονδύλια προβλέπονται για το Ταμείο Υποδεμών Connecting Euro. 336 δις προορίζονται για αυτό το ταμείο. Ε, κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι λιγότερα χρήματα από ό,τι στην προηγούμενη ε, θητεία, στην τέταρτη περίοδο. 19 δισεκατομμύρια ευρώ ή 19% λιγότερα. Ως υπερασπιστής των στόχων της περιφερειακής πολιτικής, εγώ θα ήθελα να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια και η πολιτική μας θέλει να βασίσει τις ε, να περιορίσει τις δαπάνες της ε, περιφερικής πολιτικής σε ένα ποσοστό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 231 ε, δις θα δοθούν για τη σύγκληση καθώς και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό είναι περίπου 70% του συνόλου των κονδυλίων και θεωρώ ότι έχει Ε, Το Ταμείο Συνοχής ε, θα λάβει 69 δις και για τα νέα μέλη ε, με εξαίρεση την Κύπρο και την Πορτογαλία θα πέφτει στη διάθεση των νέων μελών με εξαίρεση την Κύπρο και την Πορτογαλία αλλά χρειαζόμαστε και εδώ ένα facing out οι περιοχές που θα φύγουν από τη σύγκληση ε, χρειάζονται μία υποστήριξη της τάξης του δύο, των 2 τρίτων των κονδυλίων που λάμβαναν μέχρι τώρα. Όλες οι περιφέρειες οι οποίες ε, πρικοδοτούνται στο πλαίσιο των, ε, της σύγκλησης και όπου το ΑΕΠ είναι, υπερβαίνει το 75% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το δίκτυο και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα κατηγορία για μεταβατικές ε, περιφέρειες. Από αυτές τις περιφέρειες, από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιφελθούν εκείνες οι περιφέρειες ε, άρα συνολικά έχουμε 930 δισεκατομμύρια ε, ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ε, σας ε, περιέγραψα την παλαιά διάφρωση. Δεν υπάρχει ανάγκη για μια νέα ταξινόμηση των περιφερειών για νέες περιφέρειες που δεν λαμβάνουν κάποια χρήματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων σύγκλησης. κάθε μέτρο πρόθεσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε, ορισμένο, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Περιφέρειες με ειδικά προβλήματα θα πρέπει να υποστηριχθούν με κονδύλια που προορίζονται για τις χώρες μέλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο να προβλέψουμε ένα νέο επίπεδο χρηματοδότησης. Κατά την άποψή μου, τα κονδύλια θα πρέπει να διανεμηθούν ε, καλύτερα σε, άλλες, σε άλλους τομείς. Όλες οι υπόλοιπες ε, περιφέρειες, οι ανταγωνιστικές περιφέρειες παραμένουν και στη νέα περίοδο ε, ε, μπορούν και στη νέα περίοδο να ενισχυθούν όσον αφορά την επίτευξη των στόχων απασχόλησης. Και όλα αυτά ανταποκρίνονται στις παλιές δοκιμασμένες δομές. Για την επίτευξη του στόχου της περιφερειακής συνεργασίας υπάρχουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διατίθενται και για την πρόθεση των απομακρυσμένων περιοχών ένα δις, προβλέπεται ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Επιτρέψατε μου τώρα να σας πω κάποια πράγματα από την καθημερινή πρακτική. Μέχρι τώρα είχαμε τη ρύθμιση βάσει της οποίας ένα χάσμα μεταξύ δύο περιφερειών δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο από 20% γιατί οι περιφέρειες βρίσκονται πάντως σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους και αυτό είναι επιθυμητό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ αυτός ο κανόνας του 20% να επιδέχεται κάποιων βελτιώσεων. Ακόμα και για ένα 15% θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση για τις μειονεκτούσες ε, περιφέρειες γιατί εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο η βιομηχανία θα μεταφέρεται από τη μία χώρα στην άλλη και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ισόφελος μιας ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, κύριε, ε, ο κύριος Χάν ε, προηγουμένως μας επεσήμανε το πώς μπορεί να διαμορφωθεί, πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί μελλοντικά η πολιτική συνοχή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω ρητά την πρόθεση της Επιτροπής να προσαρμοστεί η πολιτική συνοχή στους στόχους της Ευρώπης 2020 και έτσι να προθεθούν. Ε, έξυπνα και βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα ανάπτυξης. Αυτός ο στόχος ε, διατυπώνεται τόσο για τις λιγότερο προηγμένες χώρες όσο και για τις ε, πιο ισχυρές οικονομικά περιφέρειες της Ευρώπης. Εγώ όπως και η Επιτροπή έχω την άποψη ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2013 σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να συνεχιστεί και ε, ακούμε ότι θα πρέπει να διατυπωθούν κάποιε προτεραιότητε στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά τι επενδύσει που να μπορούν να περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνεχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άπτυξη της Υπέθρου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία κλπ. Ε, όλα αυτά τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία στα οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος προηγουμένως. Η κάθε χώρα μέλος θα πρέπει στη συνέχεια να χαράξει, να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία να διατυπώνεται γραπτά σε μια ε, σύμβαση σύναψη εταιρική σχέση. Και αυτό το οποίο συμφωνείτε θα πρέπει να ελέγχεται σε αιτήσια βάση. Αυτή η στρατηγική ανάπτυξη θα πρέπει να διαφοροποιείται μέσω ενό ε, επιχειρησιακού ε, προγράμματο λειτουργικού προγράμματος. Τίποτα κυρίες και κύριοι δεν θα ήταν χειρότερο από το να σπαταλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπαθήσει κάποιους πόρους ή να τους προορίσει σε λάθος στόχους. Γι' αυτό θα πρέπει τα προγράμματα να ελέγχονται επακριβώς ως προς το περιεχόμενό τους, ώστε οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να είναι βέβαιοι ότι τα χρήματά τους δαπανώνται για τους σωστούς στόχους. Αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά τη μελλοντική συγκατάθεση των Ευρωπαίων πολιτών για την Ευρώπη, για την αποδοχή της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η Γερμανία ε, έχει μια ομοσπονδιακή διάθρωση. Ο ρόλος των διαφόρων ομόσπονδων κρατηδίων ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτές τις ε, συνθήκες. Το σύνταγμα, στο σύνταγμα, το σύνταγμα της δικής μας χώρας βάζει ορισμένου όρους και όσον αφορά την συγκέντρωση, την θεματική συνένωση των ε, σκοπών της πολιτικής, των στόχων της πολιτικής συνοχής ε, θα πρέπει ε, να συσχετιστούν με τους στόχους της Ευρώπης 2020. Για τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες, θέματα όπως ανώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αποτελούν το ένα πέμπτο των επενδύσεων, ταυτόχρονα με την αύξηση των αγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και της πρόθεσης των καινοτομιών. Ε, ο κύριος Χάν αναφέρθηκε σχετικά, η σύγκλησης και ε, θα πρέπει να βελτιώσουν τις ε, διαχειριστικές τους ικανότητες. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν ωστόσο περιφερικά προσαρμοσμένα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στο στόχο της δημιουργίας ίσων συνθήκων διαβίωσης όλων των πολιτών των ευρωπαϊκών περιφερειών. όσον αφορά τις ε, υποδομές και τη βοήθεια όσον αφορά τις υποδομές ορισμένων περιφερειών, ε, πρέπει να σας πω ότι εμείς στη Γερμανία αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε ε, να εξακολουθήσει ο συνδυασμός των τοπικών, εθνικών κονδυλίων και των κοινοτικών κονδυλίων. Εκτιμώ ότι ο Επίτροπος Χάν θα επανέλθει στο θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο. Υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση από το κοινωνικό ταμείο. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα ποσοστά τα οποία δόθηκαν. Τώρα, για να αυξήσουμε την απόδοση των ταμείων, πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα αποθεματικό 5%. Πρέπει επίσης να είμαστε πιο προσεκτικοί στην επιλογή των έργων. Από εκεί πέρα υπάρχουν και έργα, προγράμματα τα οποία ενέχουν από τη φύση τους είναι τα πιο καινοτόμα προγράμματα. Αυτά έχω τουλάχιστον στο μυαλό μου. Από εκεί πέρα το μας είπατε για την προσοχή προγραμματική περίοδο είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχω συγκεκριμένες παρατηρήσεις, υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε. Και πιστεύω ότι δεν είμαι ο μόνος που ζητά κάποιες βελτιώσεις, ολόκληρη η Γερμανία είναι μαζί μου. Οπότε, κύριε Επιτροπέ, κυρία Πρόεδρε, περιμένω με ανυπομονησία να δω πώς εσείς, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορέσετε να τροποποιήσετε το τρόπο που έχει πάρει Μέχρι στιγμής τα περισσότερα έχουν πάει καλά, αλλά όπως ξέρουμε και όπως Λέμε συνήθως ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Περιμένουμε λοιπόν επιμέρους βελτιώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε άνοδο του επίπεδου ζωής στις περιφερειές μας. Με στόχο καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και λιγότερες διαφορές, λιγότερες ανισότητες. Από την άλλη μεριά είμαστε στη διαθεσία για να μελετήσουμε περαιτέρω τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σχέντσκιν. Είναι η επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών και Τεχνολογίας. Και τώρα, από τη Βουλή της Ουγγαρίας, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Κυρίες και κύριοι, για την Ουγγαρία η πολιτική συνοχή μεταξύ των ιδιαίτερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Όχι μόνο επειδή έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο από τα κονδύλια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε καλύτερα στην περαιτέρω, περισσότερο περαιτέρω οικοδόμηση της Ευρώπης. Ε, ένας βασικός μας σκοπός είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η, ε, η Ουγγαρία ε, έχει 2,2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και 2% της ευρωπαϊκής επικράτειας αλλά τώρα έχουμε 2,7% των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας βασικός κανόνας της εφαρμογής αυτών των κονδυλίων είναι να μην υποκαθιστούν τα δημόσια έργα, αλλά να συμπληρώνονται μέσω των δημοσίων έργων και ιδιωτικών κονδυλίων. Εγώ ως βουλευτής του Ουγγρικού Κοινοβουλίου μπορώ να σας πω με περηφάνεια ότι από το 2007 έχουν δει το φως 300 προγράμματα ε, ε, της ε, τάξης μεγέθους των 38 δις. Για παράδειγμα το βιομηχανικό πάρκο, η ε, δημιουργία του πανεπιστημίου ή το σύστημα συλλογής βρόχινων όμβριων υδάτων. Είναι σκοπός μας στην Ουγγαρία να προωθήσουμε περαιτέρω την περιφερειακή πολιτική, γιατί πραγματικά η πολιτική αυτή μπορεί να εγγυηθεί μια οικονομική μεγέθυνση μελλοντικά προσδοκούμε μια ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, ούτε ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Ε, ζητούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας στον ε, παγκόσμιο ανταγωνισμό, να γίνει η Ευρώπη διεθνώς πιο ανταγωνιστική. Ε, η περιφερειακή πρόθεση θα πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης η αρχή της συνοχής θα πρέπει να διατηρήσει την πλήρη της ε, σημασία. Δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τους στόχους της Ευρώπης 2020 γιατί η συνοχή είναι εγγυήτρια της παγκοσμίου ε, ανταγωνιστικότητας. Και υπάρχει πλατεία συνένεση στις χώρες μέλη ότι η, συνοχή, ότι πολιτική συνοχή είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό ε, ε, θα πρέπει, το πνεύμα αυτό θα πρέπει να καθορίσει τις μελλοντικές συζητήσεις για την οικονομική πολιτική. Η πρόταση της Επιτροπής ε, για τους, ε, τη νέα της ε, πολιτικής συνοχής δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των φτωχότερων περιφερειών. Γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δίκαιο και παραμένει σημαντικό η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μειωθεί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Ιουνίου θεωρεί τα κονδύλια πρόθεσης των ενίσχυση των περιφερειών ε, θεωρεί τα κονδύλια ενίσχυση των περιφερειών πρέπει να παραμείνουν στο παλαιό, στα παλά επίπεδα. Αλλά αυτό δεν επιφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τις πιο φτωχές περιοχές. Και θεωρούμε ότι η επίτευξη της εδαφικής συνοχής ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πραγματικούς πόρους, πραγματικά κονδύλια. Ε, μόνο έτσι μπορούν να επενδύσουν εκεί και επιχειρήσεις των παλαιών χωρών ε, μελών. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Δηλαδή ενισχυόμενη εκ των έντων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών ε, δομών. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολλές προτάσεις που όμως περιορίζουν το περιθώριο ελιγμών των χωρών μελών. Και εδώ η Ουγγαρία έχει την άποψη θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να εφαρμόζουν όπως θέλουν τα κονδύλια της συνοχής. Για παράδειγμα, ο ΦΠΑ ε, θα πρέπει, η διαμόρφωση συντελεστή του φόρου θέμενης αξίας. Ε, δεν θα πρέπει η πολιτική αυτή να επιβαρύνει την ε, κοινοτική πολιτική. Το, η δεσμευτική δέσμη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η διαχείριση των λογαριασμών γίνεται πολύ αυστηρότερη και αυτό περιορίζει το περιθώριο ευελιξία των χωρών μελών, που όμω κατά την άποψή μου είναι σημαντική, γιατί μόνο σε ένα ευέλικτο περιβάλλον μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Τώρα, όσον αφορά του στόχου της, Ευρώπη, της Ευρώπη 2020, οι περιφέρειε ασφαλώ θα διαδραματίσουν εδώ ένα ρόλο κλειδί, αλλά όλα εξαρτώνται από τι δυνατότητε ε, και το δυναμικό των περιφερειών. Ω γενικός κανόνα θα πρέπει να ισχύει ε, ο προσανατολισμός της ε, πολιτικής προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Στις πιο προηγμένες περιφέρειες ε, θα πρέπει να παραμείνει ο στόχος προώθησης της έρευνας και της τεχνολογίας και τον τομέα εκείνων της τεχνολογίας που παράγουν προσθέμενη αξία. Ε, κατά την ε, διανομή των κονδυλίων των ταμείων θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμός, ο οποίος όμως να είναι αρκετά ευέλικτο για να ανταποκρίνεται στις ε, τοπικές, περιφερειακέ περιφερειακές ανάγκες. Μόνο μια τέτοια ολοκληρωμένη στρατηγική μπορεί να βελτιώσει τον ρυθμό μεταξύ των διαφόρων ε, ταμείων. Και ω ε, δήμαρχος προτείνω η υλοποίηση τη εδαφική συνοχή να λαμβάνει πάντοτε υπόψη της τις ε, τοπικές ε, ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες. Η εδαφική ατζέντα 2020, ε, Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει αυτή τη στοχοθεσία. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση την ολοκληρωμένη προσέγγιση για στερνιστή και Ουγγρική Προεδρία, η οποία είπε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αφού είναι ολοκληρωμένη και μόνον με τον τρόπο αυτό ε, μπορούν να βελτιωθούν οι περιφερειακοί στόχοι. Ε, συχνά ε, είναι συχνά θα πρέπει η πολιτική συνοχής να λαμβάνει υπόψη της τις λειτουργικές ανάγκες καθώς και να κινητοποιεί τις περιφερειακές και τοπικές δυνατότητες. Τα επιμέρους ταμεία δεν είναι δυνατόν να κινητοποιούνται βάσει μια ίδια λογική. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πολιτική συνοχής και τα κονδύλια της περιφερικής ανάπτυξης να έχουν ένα καλύτερο συντονισμό. Το κείμενο Αδαφική Ατζέντα 2020 ε, ψηφίστηκε στο Γκούντουλε από τους αρμόδιους υπουργούς. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει πολλούς στόχους μια ισορροπημένη ανάπτυξη, μια βελτίωση της σχέσης μεταξύ ε, πόλων και υπαίθρου, ε, διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων εδαφικών περιοχών, ε, οικολογία και πολιτιστικές αξίες. Υπό το πρίσμα αυτό θεωρώ σημαντικό το διοικητικό άχθος κατά τη διανομή των κονδυλίων να μειωθεί γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια όσον αφορά, τόσο όσον αφορά τους αποδέκτες όσο και τις χώρες μέλη. Επειδή η αποτελεσματικότητα των επιμέρους προγραμμάτων εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή, η λύση δεν μπορεί να είναι η αύξηση των διοικητικών εμποδίων, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, το σκεπτικό. Δηλαδή το ζητούμενο είναι οι μηχανισμοί εκτέλεσης της πολιτικής συνοχής να διαμορφωθούν με πιο διαφανή τρόπο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν τα ποσοστά σφάλματος. Είναι σημαντικό ήδη πριν από το 2014 να θεσπίσουμε μια ξεκάθαρη δέσμη κανόνων. Θεωρώ ότι παραμένει σημαντικό τα κονδύλια μελλοντικά να μπορούν να χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο και τα αποτελέσματα και τα, και τα αποτελέσματα να ελέγχονται ήδη και να προγραμματίζονται εκ των προτέρων. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω πολιτική συνοχή να παραμείνει σημαντικό επίτευγμα της ευρωπαϊκής πολιτικής και μετά το 2013 να μην χάσει δηλαδή την βαρύτητά της. Ως εκπρόσωπος μιας κοινότητας, μιας ε, πόλης της Υπέθρου θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου οι αρμόδιοι πολιτικοί να φερθούν ε, με νοήμονα τρόπο και προς εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος και να συμφωνήσουν επί των κοινών κανόνων. Uh, our next speaker is Mr. Vili Ο κύριος Βαλή Τροφενίκ από τη Σλοβενία είναι ο επόμενος ομιλητής επικεφαλής της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί προσκεκλωμένοι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τις δικές μας προτάσεις και απόψεις επί της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστειλε ΦΕΣ μήνυμα περί αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών μας και έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη, να πετύχει προσθεμένη αξία, να διευκολύνει τον εξυγχρονισμό, και την αηφόρο ανάπτυξη. Είναι όμω πρωταρχικός μήνυμα αλληλεγγύης. Από εκεί πέρα για την ε, μεταβολή του κλίματος, για την ανταγωνιστικότητα, την παγκοσμιοποίηση κλπ. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει. Όλα αυτά εντός του δημοσιονομικού πλαισίου. Ταυτόχρονα δεν ξεχνώ ότι υφιστάμεθα κρίση δημοσιονομική κάτι το οποίο μειώνει τα περιθώρια λιγμών για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τους εθνικούς όσο και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπό την άποψη αυτή, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ρεαλιστικό. Προβλέπει σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών και περιέχει μέτρα για την ε, αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σημειώστε πάντως ότι ο περιορισμένος κοινωτικός προπολισμός μπορεί να μας αφήσει να προχωρήσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε επιπλέον θέσεις εργασίας. Και αυτό γιατί όλα αυτά συνδέονται με την στρατηγική 2020. Χρειαζόμαστε προφανώς έναν ικανό προϋπολογισμό για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Τα κονδύλια είναι η μόχλευση για την δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας. Από αυτήν την άποψη, η πολιτική συνοχής και το πολιτές πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του 2020. Συνεπώ, η συνοχή πρέπει να συνεχίσει να είναι παρούσα στον κοινωνικό προπολισμό. Και αυτό το λέω όχι μόνο για την ανάπτυξη και τις θέσει εργασία, αλλά και διότι εργαλείο έχει ήδη δοκιμαστεί με καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση. Η πολυεπίπεδη αυτοδιοίκηση, η τοπική και η περιφερειακή, επίσης δούμε προς το συμπέρασμα αυτό. Ανεξαρτήτως των προσπαθειών που ήδη καταβάλουμε στην πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί μας δεν θα είναι επαρκείς ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση για την κάλυψη των απαιτουμένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και απαιτητικοί. Η πολιτική συνοχής θα κινητοποιήσει πόρους στα μία από τις βασικές πολιτικές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε σύγκληση είναι πολιτική συνοχή. Εννοείται ότι οι περισσότεροι πόροι πρέπει να απορροφηθούν από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό είναι και ελληνική άλλωστε. Έτσι θα ενισχύσουμε αυτό που ονομάζουμε συνοχή. Η πολιτική συνοχή πάντως πρέπει να είναι παρούσα παντού γιατί όχι μόνο θα ενισχύσουμε παντού την ανταγωνιστικότητα για να πετύχουμε τους στόχους της κάθε περιοχής. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε μια συνέχεια στην χρηματοδότηση της μιας ή της άλλης περιοχής, χωρίς εκπλήξεις και απότομες αλλαγές. Η κρίση, είναι η κριση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις περιφερειές μας. Η κρίση μπορεί να καταστρέψει τις προοπτικές ανάπτυξης μιας περιφέρειας, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και τις σημερινές. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκείς μηχανισμούς μετάβασης, όπου και το λεγόμενο phasing out θα γίνει με τρόπο σταδιακό. Οι χώρες δηλαδή που έπαιρνε χρήματα μέχρι το 2007 όντα πάνω το 50% του κατοικοφέλην ΑΕΠ, θα έχουν και αυτέ κάποια στήριξη. Τώρα, όσον αφορά την κατανομή μεταξύ χωρών. Γενικώ συμφωνούμε. Όμω τα 10 δι για το Connecting Europe μου φαίνεται λίγο παράδοξο. Είπαμε να εξελίξουμε εμπόδια, αλλά τα σημερινά εμπόδια, θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε με μια κεντρική ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με αυτό λοιπόν διαφωνώ με τα 10 δισεκατομμύρια για το Connecting Europe και σε κάθε περίπτωση ζητώ να γίνουν σεβαστά τα λόγω κριτήρια. Και αυτό θα πετύσει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν κάθε φορά που θα προκρίνονται προγράμματα προτεραιότητας. Κάτι άλλο. Τα σχέδια εδαφικής συνοχής. Αυτά διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων καθώς και τη συνεργασία με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτό είναι και, το, και η αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ενισχύουμε προγράμματα μεταξύ άλλων διασυνοριακής συνεργασίας. Πολλές φορές αυτά είναι προγράμματα εξαιρετικά σημαντικά για τις πλέον απομεμακρυσμένες περιοχές. Αναπτύσσοντας σχέσεις, ενισχύουμε και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή όμως πρέπει να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό καθιστά μια πολιτική χρήσιμη. Οι λεγόμενες λοιπόν αιρεσιμότητες εδώ, εν είναι χρήσιμες. Έχουμε και υποχρεώσεις όμως, όπως η Agenda του 2020. Έχουμε τα εθνικά προγράμματα. Και αυτό είναι καλό. Γιατί όλα αυτά θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα προκύψουν έτσι νέες δομές στην αγορά και στην αγορά εργασίας. Έχω από την άλλη μεριά τις αμφιβολίες μου όσον αφορά την χρησιμότητα των κυρώσεων γιατί αυτό σίγουρα δεν αποτελεί ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών. Δεν είναι δημοκρατικός αυτός ο κανόνας ούτε οδηγεί καλά αποτελέσματα. Οπότε περνάμε στην λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα τους κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις ένα μακροεπίπεδο. Στόχος των προσπαθειών, όπως ε, προείπα, είναι να έχουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Με προκειμένου κάποια κρατημέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες του χωριούνται κονδύλια και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Εμεί πρέπει παρ' αυτά, μάλλον και γι' αυτό τον λόγο, να θέσουμε συγκεκριμένε προποθέσει, απαιτήσει και κριτήρια πριν εγκριθεί ένα κονδύλι. Έτσι, περιφέρειες, ε, νομοί, κράτη θα πρέπει να σκέφτονται και να αναλύουν πριν κάνουν την οποιαδήποτε αίτηση. Φυσικά την πολιτική αυτή δεν πρέπει να την ε, φορτίσουμε, δεν πρέπει να την επιβαρύνουμε με τις επιμέρους σκέψεις του ένας και του άλλου. Αυτό θα καταλήξει μια κακή πολιτική συνοχή, ενώ τώρα αποδίδει. Έχει ευνοήσει τις επιχειρήσεις, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. κλπ. Οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, απλή και κατανοητή. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ως προς τους κανόνες, το πλαίσιο μας να τροποποιηθεί. Πρέπει να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τον αριθμό των φορέων, ειδικά των, των ελεγκτικών φορέων που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και να εφαρμόσουμε μια πιο πρακτική πολιτική προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εντός των οποίων θα έχουμε και θεματικές προτεραιότητες. Αυτό όμως μας παρέχει περισσότερη ευελιξία, είναι πιο εύκολο. Οπότε, αυτό με φέρνει στις δημόσιες συμβάσεις, στον κανόνα νησιν 2, όπως γνωρίζετε, περιφέρειες ασχολούνται συνήθως με το να βρουν τα κονδύλια και όχι με το πώ θα τα Αυτό είναι σχεδόν φιλοσοφικό θέμα, διότι για άλλε αναπτυξιακέ πολιτικέ πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, τι κάνει το ΕΤΠΑ. Τι γίνεται με την επικουρικότητα. Τι γίνεται με τα σύμφωνα Εταιρική σύμπραξη. Χρειάζεται σίγουρα στρατηγική εμπλοκή σε αυτά τα θέματα και σύμπηξη συμμαχιών. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε τα κείμενα αυτά, τα μέτρα αυτά να μην αυξήσουν το βάρος για τον προπολογισμό. Μία προϋπόθεση για την δρομολόγηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 είναι η έγκυρη κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το προσεχές πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών. Κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μέσα στου επόμενου 18 μήνες. Είμαι βέβαιος ότι το εθνικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν προκειμένου να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Τροφένικ. Τώρα θα προχωρήσουμε στους επόμενους αγορητές που δεν θα έχουν όμως τόσο χρόνο στη διάθεσή τους. Έχουμε 15 εγγεγραμμένους ομιλητές για την ώρα. Μπορώ να δώσω 4 το πολύ 5 ε, λεπτά ομιλίας για τον κάθε έναν, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προσταθούν και άλλοι στον κατάλογο αυτό. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπη, αγαπητοί εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί συνάδελφοι. Με την έναρξη σήμερα της διαδικασίας για την υιοθέτηση του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής συνοχής, πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ευθύνη μα είναι να επικεντρωθούμε στα αδύνατα σημεία τη πολιτική προκειμένου να βελτιώσουμε και όχι να θέσουμε νέα εμπόδια στην υλοποίησή τη. Καλωσορίζουμε τι περισσότερε από τι προτάσει τη Επιτροπή, οι οποίε αποτελούν άλλωστε και τι κύριε θέσει του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον τη πολιτική, όπω τη στήριξη πολλών ε, όλων των περιφερειών, η δημιουργία μια ενδιάμεση κατηγορία στήριξη, η επικέντρωση στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, η προσπάθεια απλοποίηση των κανόνων και τη διαχείριση, η αναλογικότητα στους ελέγχους. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ σε ένα σημείο για το οποίο κατ' επανάληψη και μέσα από πολλά ψηφίσματα έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή μας. Καταρχήν δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί την ανάγκη για πιο ποιοτικά και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχων και αξιολογήσεων και για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής περισσότερο προσανατολισμένης στα αποτελέσματα. Στις βασικές, στις σχετικές διαβουλεύσεις, ωστόσο, πάνω στις οποίες βασίζονται οι σημερινές προτάσεις, η πλειοψηφία των φορέων τάχθηκε κατά της εισαγωγής προϋποθέσεων, τις οποίες οι ίδιοι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση φορείς δεν μπορούν να ελέγξουν. Είναι οι γνωστές μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε έγγραφο της ίδιας της Επιτροπής αναφορικά με τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων επί της πέμπτης έκθεσης για τη συλλογή. Θα φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να τιμωρούμε τις περιφέρειες για πολιτικές προϋποθέσεις και λάθη τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ελέγξουν και για τα οποία συνεχώς δεν φέρουν την ευθύνη. Ω Κοινοβούλιο έχουμε εκφράσει με σχετικά ψηφίσματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί με συντριπτική πλειοψηφία την αντίθεσή μα στην εισαγωγή οποιονδήποτε προποθέσεων που δεν σχετίζονται με την ίδια την πολιτική και του στόχου τη. Για να είμαι ειλικρινή, πίστευα ότι η θέση τη Επιτροπή κινείται στο ίδιο πνεύμα. Αλλά οι σημερινέ προτάσει αποδεικνύουν το αντίθετο. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή πώς φαίνεται τελικά, πώς φτάσαμε τελικά στη σημερινή πρόταση η οποία συνδέει και μάλιστα κατά πολύ άμεσο τρόπο τη χρηματοδότηση μέσων των ταμείων της πολιτικής συνοχής με τις μακροοικονομικές πολιτικές του κάθε κράτους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής, ώστε να αποτελέσει αυτή μια ισχυρή βάση που θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού κάθε περιφέρειας και θα εγγυάται τη συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ενώ είπα προηγουμένως ότι ο καθένας θα μιλάει 4-5 λεπτά, προστέθηκαν άλλοι 10-15 ε, αγορητές, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος. Ιωάννα Βόσα από τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Θα εκφραστώ σύντομα. Εν ώψη των απαιτήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διατυπωθεί πάρα πολλά προβλήματα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσέγγιση της Κομισιόν. Αυτό αφορά τη διατύπωση προτεραιοτήτων και τη διασύνδεση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ευρώπη ε, προγραμματίζει ένα κατάλογο με προτεραιότητες που λέει πού θα πρέπει να προορίζονται μελλοντικά τα κονδύλια της Ένωσης. Και αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να προσανατολίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Και μια τέτοιου είδους διασύνδεση είναι προβληματική κατά την άποψή μας. Γιατί οι περιφέρειες κατά την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν έχουν τη διαθέσιμη, την αναγκαία συγγνώμη, ευελιξία. Άρα λοιπόν η βάση της πολιτικής συνοχής που είναι ο συγκεκριμένος προσανατολισμός προς τις συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειών χάνεται. Ε, το Ταμείο Αλίας ή το Ταμείο Ανάπτυξης Υπέθρου ε, έχει κάθε ενδιαφέρον για μια ενίσχυση της πολιτικής συνοχής η οποία δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα ε, εκφυλισμένο εργαλείο εκτέλεσης της, προ... πολιτικής για την εφαρμογή της Αττικής Ευρώπη 2020. Αυτό ισχύει ιδιαίτερος για το EFS η Κομισιόν προγραμματίζει την εκταμείευση κάποιων κονδυλίων εξαρτώντας την από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στις χώρες μέλη. Και στο επίπεδο χωρών μελών ε, οι αποφάσεις θα ληφθούν χωρίς συμμετοχή των περιφερειών. Με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τον αρχικό στόχο, δηλαδή την ε, μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό απορρίπτουμε τέτοιου είδους ε, ε, ρεσιμότητα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο δημιουργούνται κάποιες εταιρικές σχέσεις χωρίς να αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, απορρίπτουμε αυτού του είδους την πολιτική που αποκλείει τις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ματσόνη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια ε, για την ταχύτητα με την οποία οργανώσατε αυτήν την ε, ακρόαση, συζήτηση για την ε, πολιτική συνοχής. Εγώ εξετίμησα ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα πράγματα η Πολωνίδα υπουργό και ελπίζω ότι θα υπάρξουν οι συνθήκες οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα ε, πολύ γρήγορα ε, να υλοποιηθούν τα πράγματα όπως έγινε και στις, προηγου... στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κ. Χάν για τον τρόπο με τον οποίο ε, ανάγλυφα παρουσίασε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως θα χρειαστούν τι να εμβαθύνομαι. Θα ήθελα εξ αρχής να κάνω κάποιες πάρα πολύ γρήγορες σκέψεις. Πιστεύω ότι η πρόταση που μας έχει υποβληθεί ε, είναι συνεκτική με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει ε, με την ε, υλοποίηση του στρατηγικού πολιτικού του οράματος, ε, γιατί πλέον οικοδομείται ε, σε στενή συνεργασία με τους στόχους της στρατηγικής 2020 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, παρόλα αυτά, δεν καλύπτουν οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά συγκεκριμένες στοχευμένες προτάσεις για απλούστευση, συγκέντρωση και στοχοπροσύλωση ε, και προσήλωση στα αποτελέσματα, πράγμα που επανειλημμένα έχουμε εκδηλώσει εμείς ε, σαν Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά μας. Ε, πιστεύουμε ότι δεν παράγεται απαραίτητα απλούστευση, η μείωση των προγραμμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα συγκέντρωση στους στόχους και επομένως όχι απαραίτητα στόχοι οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για την νέα Ευρώπη 2020. 20 και ότι καμιά φορά και η αιρεσιμότητα ε, κρίνεται από, με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Επίσης να πω ότι το όραμα έτσι όπως αυτό ε, αναδύεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μερικές φορές ε, κινδυνεύει να προδώσει τον ίδιο του το στόχο, δηλαδή ε, να λάβει υπόψη τις ε, εδαφικές, γεωγραφικές πραγματικότητες ε, των πιο μειονεκτικών περιοχών. Θετικό πρόσημο βεβαίως βάζουμε στο βάρος το οποίο έχει δοθεί στην εδαφική διάσταση, στο, στα πλαίσια της νέας στρατηγικής, κυρίως δε για την ιδιαίτερη υπογράμμιση που δίνεται ε, στην αστική ατζέντα. Ε, λείπει όμως ε, η διασύνδεση με τις υποαστικές περιοχές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως θα είναι και πάρα πολύ σημαντικός ο ειδικός τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί τι ε, το θέμα του επιχειρηματικού ιστού, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς όλα αυτά τα μέτρα ε, θα μπορέσουν να ε, ωφελήσουν τελικά όλους αυτούς τους συμμετέχοντες στην πολιτική συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω ε, κάποιες, ε, ε, κάποιους δισταγμούς όσον αφορά την αιρεσιμότητα εξπόστη και εξάντε και σε διασύνδεση με τις μακροοικονομικές επιλογές. Βεβαίως εγώ συμφωνώ με την βελτιωμένη εξάντε αιρεσιμότητα που δίνει την δυνατότητα τα προληπτικών δράσεων όσον αφορά την υλοποίηση των ε, σχεδίων και βεβαίως ε, συμφωνούμε και με την αιρεσιμότητα βάση αποτελεσμάτων αν και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να οριστεί με καλύτερο τρόπο. Όσον αφορά τώρα τις διαφορετικές αιρεσιμότητες ε, που ε, βασίζονται σε εθνικές παρεμβάσεις, σε παρεμβάσεις από των κρατών μελών, ε, εδώ δεν είμαστε απολύτως συμφωνοί, γιατί εδώ ο χρόνος που χρειάζεται πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερος από, τον, από τα χρονικά όρια τα οποία προβλέπονται στην πρόταση. Πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια αιρεσιμότητα δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ε, πολιτική την οποία θέλουμε εμείς και επίσης δεν είναι δυνατόν η οικονομική πολιτική να τραβήξει ε, την ε, περιφερειακή πολιτική την πολιτική συνοχής πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα προγράμματα σταθερότητας βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αλλά δεν είναι δυνατόν ε, να αποτελέσουν παράθερα πενίδες της ε, κύριας ε, περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής. Στη, για τις μεταβατικές περιοχές τώρα βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, καθοριστούν οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι κατά προσέγγιση. Ε, η εισαγωγή αυτή δεν πιστεύουμε ότι θα φέρει συνολικά ωφέλη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε δεν ευθυγραμμίζεται με το ίδιο το πνεύμα της πολιτικής συνοχής. Ιδίω δε τα στοιχεία τα οποία διαβάσαμε και τα οποία αντιμετωπίσαμε μας οδηγούν ε, στο ε, να πούμε ότι εάν 70 εκατομμύρια ε, πολίτες Ευρώπης ίσως, ίσως θα μπορέσουν να ωφεληθούν, δεν είμαστε σίγουροι από αυτό το νέο στοιχείο, οπωσδήποτε θα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός για τον πολιτών εννοείται, ε, για τους οποίους θα προκύψει ζημία και επομένως το σημείο αυτό ουδόλως ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις που είχε κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να πρέπει να μπουν σε ένα ε, ε, ενιαίο πρόγραμμα και επομένως ε, δεν νομίζω <coughs> ότι βλέπουμε να υπάρχει συγκέντρωση πόρων. Ένα, ένα τελευταίο αίτημα αποσαφήνισης αφορά το Ταμείο Συνοχής, το οποίο αλλάζει τους κανόνες του, <coughs> χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται σαφώς τι θα γίνει ε, ε, όσον αφορά τον καθορισμό των πόρων που θα έχουμε στην διάθεσή μας. Επίσης, χρήση ενός τμήματος του Ταμείου Συνοχής ε, για την πολιτική διασύνδεση της Ευρώπης, καθώς επίσης και η ιδιαιτερότητα του Ταμείου Συνοχής που μας δημιουργούν προβληματισμούς και δισταγμούς όσον αφορά την δυνατότητα υλοποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε τρία λεπτά η κυρία Άντζελα, <laughs> Γκερέκο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ευτυχής που έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε μια τόσο σημαντική συνάντηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Είναι σαφές ότι ένας από τους κεντρικούς άξονες του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Προερχόμενη από μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με δεδομένες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, οφείλω να επισημάνω ότι το πρόβλημα της πρημοδότησης των δυσπρόσωτων περιφερειών ή και περιοχών για μας είναι κρίσιμο. Αναμφίβολα η νησιωτικότητα μιας περιοχής είναι επιβαρυντικός παράγοντας σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητά της. Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα των μεταφορών και των συγκοινωνιών είναι απολύτως κρίσιμο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και την περαιτέρω επίτευξη συνοχής. Κατά συνέπεια θεωρώ πως πολιτικές όπως αυτή του μεταφορικού ισοδύναμου οφείλουν να αποκτήσουν πρωταρχικό χαρακτήρα προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι όπου έχει αξιοποιηθεί έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Ειδικά για το θέμα της νησιωτικότητας, η επιλογή μιας οριζόντιας πολιτικής για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης είναι μια λύση. Δεδομένου ότι το πρόβλημα προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά και άλλες περιοχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση της Επιτροπής που έχει κατατεθεί στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 28 και 29 Ιουλίου στην Πολωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία ταμείου για τις υποδομές, ενώ καταρχήν κάτι τέτοιο ακούγεται θετικό ως ιδέα, μας προβληματίζει το γεγονός ότι δημιουργείται ως νέο θεματικό ταμείο, το οποίο εκ των πραγμάτων θα εξυπηρετεί έργα σε δίκτυα όπως το TEN-T και το TEN-E, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι νησιωτικές περιοχές. Επομένως, στην πράξη το Ταμείο Υποδομών δεν θα μπορεί να θεωρεί επιλέξιμες τις περιοχές αυτές που λογικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα. Σημαντική επίση θεωρώ και την πρόταση σχετικά με τη δημιουργία της ενδιάμεσης κατηγορίας περιφερειών με βάση το ΑΕΠ Εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη δυνατότητα για να πρημοδοτηθούν οι περιοχές προβληματικής πρόσβασης, όπως αυτές που ανέφερα προηγουμένως, νησιωτικές και ορεινέ να συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη νέα ενδιάμεση κατηγορία θα θεωρούνται ως επιλέξιμες περιφέρειες με σαφείς γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως τα νησιά και οι ορεινοί όγκοι, ανεξάρτητα από το ΑΕΠ που παρουσιάζουν. Θεωρώ τέλος ότι η απλοποίηση των διαδικασιών, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οφείλει να είναι αυτονόητος στόχος του νέου προγράμματος. Νομίζω ότι είναι κοινή αποδοχή ότι υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη γραφειοκρατική πολυπλοκότητα στις διαδικασίες, η οποία μας κοστίζει πολύ σε αποτελεσματικότητα. Το θέμα φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει αυτή η δημόσια συζήτηση στα πλαίσια της συγκεκριμένη διαβούλευσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καρυματέλη. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Και το λεφτό διότι αισθάνομαι ότι αποκαθίστεται η δεσμοί με ένα παλιό εργαλείο, το Urban. Έτσι, το ΕΤΠΑ θα κάνει την παρουσία του πιο αισθητή στα μάτια και των ερετών. Έτσι, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ θα δώσουν μάχη κατά της φτώχειας και της ενεργείας. Θα αποφεληθούν έτσι οι μικρές συνοικίες των αστικών συγκροτημάτων. Μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ πρέπει να προκύψει μεγαλύτερη συνέργεια σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για την ενεργειακή απόδοση. 20% των εθνικών προϋπολογισμών από το ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το ερώτημά μου όμως είναι απλό. Υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρξει ειδικό προπολογισμό για την βελτίωση των κτηρίων και ειδικά των ε, λαϊκών κατοικιών. Πιστεύω ότι το μέτρο είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τις λαϊκές γειτονιές. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μου εγγυηθείτε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ευχαριστώ. Thank you from uh, National Rat of Austria. από την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα κύριε Επίτροπε. Εμείς στην Αυστρία φυσικά χαιρετίζουμε τις ε, προτάσεις του Επιτρόπου για την πολιτική της. Ε, γιατί με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων ενίσχυσης των περιφερειών. Η στρατηγική της ενίσχυσης ε, των ενισχύσεων έχει ε, διαμορφωθεί με πολύ πιο διαφοροποιημένο τρόπο ε, γι' αυτό κατά την άποψή μας θα μπορέσει να επιτύχει πολύ αποτελεσματικότερα τους στόχους από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Ιδιαίτερως θα ήθελα να τονίσω το εξής. Εάν ε, ο ανταγωνισμός ε, μεταξύ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ περιφερειών που λαμβάνουν ενισχύσεις και αυτών που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις. Ε, εδώ θα πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους ανισότητες. Συνολικά χαιρόμαστε για το γεγονός που μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ε, γιατί και στο παρελθόν ε, είχαμε τέτοιου είδου εργαλεία. Εάν δούμε την στρατηγική Ευρώπη 2020, διαπιστώνουμε ότι η πολιτική συνοχής και η πολιτική ενίσχυση των περιφερειών θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα είναι σημαντικό να διατυπωθούν οι προϋποθέσεις πλαίσιο ιδιαίτερως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τον τομέα των υπηρεσιών γιατί ο τομέας των υπηρεσιών έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων ε, απασχόλησης, αλλά ε, χρήση βελτιώσεων. Βλέπουμε εδώ ένα μεγάλο δυναμικό. Και οι αποδοχές ε, είναι, βρίσκονται υπό πίεση και πολύ συχνά επιφέρουν τις επιπτώσεις των, ε, της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων ε, υλών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να επενδύσουμε όλες τις προσπάθειές μας στην πρόθεση της καινοτομίας. Επίσης το θέμα της επιμόρφωσης. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να δω να συμπεριλαμβάνει τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Συνολικά είμαστε ιδιαίτερος ε, ικανοποιημένοι με τις προτάσεις του Επιτρόπου κ. Χάν. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς ε, ικανοποιημένους εδώ. Και τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και πάλι Μαρίνα Πέρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η στάση της πολιτικής μου ομάδας ε, ε, καθορίστηκε από την παρέμβαση του συνάδελφου του κυρίου Σταυρακάκη όσον αφορά τη μακροοικονομική πολιτική. Αλλά επιτρέψατε μου να πω ε, το εξή. Η προτεραιότητα είναι μεν η σταθερότητα, αλλά ε, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Αυτό είναι ο βασικό στόχο. κύριε Επίτροπε, έχω ορισμένε ερωτήσει, αλλά θα περιοριστώ σε τρει από αυτέ. Η πρώτη ε, σχετίζεται με μία σημείωση που εμφανίστηκε στον Ισπανικό τύπο. Υπάρχει μία γενική ανασφάλεια μεταξύ των πολιτών γιατί η Κομισιόν προτείνει να αναστείλει τις περιφερειακές ενισχύσεις σε ελληματικές χώρες, σε χώρες μέλημα. Ε, η Επιτροπή προτίθεται πράγματι να παγώσει τις περιφερειακές ενισχύσεις προς αυτές τις χώρες. Δεύτερον, όσον αφορά την ενδιάμεση κατηγορία, επιτρέψατε με να γίνω πιο ρητή. Μπορεί ο Επίτροπος να εξηγήσει λεπτομεριακά πώς θα υλοποιηθεί η διανομή των κονδολίων μεταξύ περιφερειών που θα συμπεριλάμβουν τη νέα ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών, ε, δηλαδή περιφέρειες που δεν επιφωνούνται πλέον από τις ε, ενισχύσεις σύγκλησης. Και η τρίτη ερώτηση αφορά το αποθεματικό αποτελεσματικότητας. Ε, η Επιτροπή θέλει να επανεισάγει αυτό το αποθεματικό παρόλο που στο παρελθόν αποδείχθηκε αποτελεσματικό και με υψηλό διοικητικό άχθος. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει το σύστημα αναθεώρησης των εσόδων να μην ε, βασίζεται σε, ε, βασίζεται σε προγράμματα, βασίζεται σε προγράμματα τα οποία έχουν την καλύτερη απόδοση από, τον, ε, από την Αυστριακή Βουλή. Κύρια Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, εξάρτημες κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Ο Κόνραντ Στάινελ ανέφερε ήδη την αυστηρική, ήδη την αυστηρική θέση ε, για την πρόταση της Επιτροπής, που την εξολογούμε πολύ θετικά. Εμείς σε αντίθεση με ορισμένου συναδέλφου από εθνικά κοινοβούλια, μπορούμε να φανταστούμε το πρόγραμμα ενίσχυση να συνδέεται με δημοσιονομικά μέτρα. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ε, μπορεί να υλοποιηθεί διορθωτική πολιτική. Δεν μπορεί βεβαίω να υποκαταστήσει ποτέ την εθνική πολιτική μπορεί να είναι μόνο ένα μέσο προώθησης της ευημερίας σε εθνικό επίπεδο. Η αυστρική τοποθέτηση είναι ανοιχτή για μια καινοτομία στη συγχρηματοδότηση ε, όσον αφορά περιφερικά δύναμες ε, περιοχές και για μας είναι, μπορούμε να φανταστούμε να μειωθεί το μερίδιο της συγχρηματοδότησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα τους, ώστε να δώσει κανείς αυτές τις μειονεκτούσες περιφέρειες τη δυνατότητα πρόσβασης αυτές τις ενισχύσεις. Για το, το διάστημα 2004-2020 θα είναι ως βάση για τα κονδύλια συνοχής και εμείς ως Αυστριακοί ε, αποβλέπουμε κυρίως την επίτευξη της διαφάνειας ε, και για τα ευρωομόλογα εντός του δημοσιονομικού πλαισίου και όχι εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου, ούτε ώστε να παρεμπεδίσουμε ε, να παρακαμφθεί η απαγόρευση της υπερχρέωσης των κρατών η οποία δράζεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Χάν για την ε, πρότασή του και θα ήθελα να πω ότι η ομάδα Άλτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις ε, απλουστεύσεις τις οποίες ζητήσαμε κατά επανάληψη, μια απλούστευση των κανόνων, μια απλούστευση της διαχείρισης επίσης. Και χαιρετίζουμε επίσης την αύξηση της οικονομικής επίδοσης ε, μέσω της, του, του προσανατολισμού των επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το ΆΛΔΕ ε, ε, ζητάνε το ίδιο και όσον αφορά το αποθεματικό. Ε, εμείς είχαμε ζητήσει πάνω από 15% για αυτό το αποθεματικό όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων και τους κοινού κανόνες που θέλουμε να επεξεργαστούμε ε, σε όλα αυτά αναφέρεται η πρόταση. Αλλά διαπιστώνουμε, και διαπιστώνουμε ότι οι χώρες μέλη συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα και σε εθνικό επίπεδο να προτείνουν κάποιους επιπλέον επιπρόσθετους κανόνες, κανόνες που είναι επιπρόσθετοι στους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συμφωνημένους κανόνες. Κάτι που θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα μία υπερπληθώρα της ρύθμισης και αυτό δεν θα ήταν τελικά εσόφελος των ε, πολιτών. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια πραγματική απλούστευση που να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Και σε συνάρτηση με αυτή την απλούστευση των κανόνων θα ήθελα να φερθώ και σε μια πρόταση της Επιτροπής. Αναφέρεται ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να μειώσουν τις ε, αρμόδιες για τη διαχείριση των ταμείων αρχέσα. Ε, είναι, η ερώτηση μου είναι κατά πόσο είναι αναγκαίο να γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή όταν προτίθενται να λάβουν τέτοια μέτρα. Δεν θεωρείτε όμως ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγεί σε κάποιες ανισορροπίες όσον αφορά την ε, διανομή των κονδυλίων. Ε, το ΆΛΔΕ συμφωνεί όσον αφορά την ερεσιμότητα, αλλά θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο που η βασική αυτή αρχή της ερεσιμότητας ε, εφαρμόζεται στην πράξη. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Κατ' επανάληψη επισημαίνεται η αξία των αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. Αλλά σε αυτό δεν αναφέρεται καθόλου η πρόταση της Επιτροπής και εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία της πολιτικής συνοχής εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τους, ε, από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες θα πρέπει επιτέλους να υλοποιήσουν την ε, πολιτική συνοχής. Όσον αφορά, τώρα, όσον αφορά την απλούστευση, η θέσπιση του μοντέλου e-cohesion, δηλαδή τα, η ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως το χαιρετίζουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας οδικός χάρτης για τις χώρες μέλη, ούτε ώστε να μπορούν να προτεμαστούν για αυτές τις ηλεκτρονικές ε, ε, δομές γιατί το 2014 θα πρέπει να λειτουργεί το σύνολο αυτού του συστήματος. Και από αυτό θα εξαρτηθεί η επιτυχία αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος ή cohesion. Ευχαριστώ κύριο καραβάλια από την ε, Ελκυή Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε ως προς τους στόχους Συμφωνούμε με την απλούστευση, την ε, απόδοση, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και συμφωνούμε να δώσουμε αγώνα για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Αυτό αφορά τι επιχειρήσει, κυρίω βεβαίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Στην ε, χώρα μου, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αντιπροσωπεύουν 85% τη απασχόληση και 70% των επενδύσεων και τη προσθεμένη αξία. Τώρα, ακριβώ επειδή μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί το πραγματικό πρόβλημα ε, αυτών των ε, μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, η πρόσβαση στην τραπεζική πίστη, που με τη Βασιλεία 3 γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και φυσικά δυσχεραίνεται και από την παρούσα κρίση. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ε, ένα ένα απλό μέτρο χρήσης ε, των ε, κονδυλίων των εθνωτικών ταμείων για τη δημιουργία ενός ταμείου εγγύησης έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην πίστη ε, και στις πιστώσεις και επομένως να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και βεβαίως τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες θα μπορούσαν να ελέγχουν την σκοπιμότητα των αναπτυξιακών ε, προγραμμάτων ε, και ακριβώς λόγω της έλλειψης ε, και των πόρων θα μπορούσαμε να καλύψουμε το πρόβλημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα, μια και ορθώς τίθεται ο στόχος της μείωσης της ανεργίας, κυρίως δε της ανεργίας των νέων, και εν προκειμένου ε, ζητούμε ε, να χρησιμοποιηθούν, ε, αν είναι δυνατόν λέω, να χρησιμοποιηθούν κάποιοι πόροι των εκδοτικών ταμείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πρόσληψη νέων ανθρώπων, βεβαίως μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο, ο κύριος Ιστερόη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, βρισκόμαστε μεταξύ φίλων, φίλων ε, και φίλων και της συνοχής ε, βέβαια. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Επίτροπος θα έχει αυτήν την αίσθηση και δεν είναι η ίδια αίσθηση που είχε με την επιστολή των οχτώ ε, χωρών, γιατί υπήρξε μια τέτοια επιστολή που έλεγε ότι αμάν πια με αυτές τις φτωχές περιοχές και τι θα γίνει πια με αυτά τα χρήματα. Ε, φυσικά πρέπει ε, να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα σε εθνικό επίπεδο και φαντάζομαι φυσικά θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια και οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις ε, και ενδεχομένως και κάποια αγκαθάκια όταν θα πρέπει ε, να ευθυγραμμίσουμε αυτές τις πολιτικές ε, με την παρούσα οικονομική κρίση, με τα μακροοικονομικά στοιχεία κτλ. Ε, όμως, όμως δεν πρέπει ε, αυτά τα οποία να λέμε εδώ να μιλάμε μονάχα για περιφερειακή πολιτική ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, εταιρικές σχέσεις ε, οι οποίες λειτουργούν πολύ καλά. Απ' την άλλη παιδιά υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στα περιφερειακά κοινοβούλια και που μας δημιουργούν κάποιο προβληματισμό. Εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι ότι συζητάμε, συναντιόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, εμβαθύνουμε. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το λέω με τα λόγου γνώσεως ε, ε, έδειξε μεγάλο θάρρος καταθέτοντας τις προτάσεις της, βάζοντας την πολιτική συνοχή στο κέντρο των μελημάτων της. Ολοκληρωμένη προσέγγιση θέλουμε εμείς και πολύ χρόνο πήρε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι να το κάνει και εκείνη. Μέχρι πριν από ένα-δύο χρόνια ε, οι πολιτικές ήταν κατακαιρματισμένες πότε για τους υδατινούς πόρους, πότε για το περιβάλλον, πότε για το ένα, πότε για το άλλο, ενώ εδώ δίνεται πραγματικά η δυνατότητα ε, ολοκληρωμένου προγράμματος, ενιαίου προγράμματος που μπορεί να ε, ε, αντιπροσωπεύσει επάξια την Ευρώπη σε έναν ε, διαρκώς κινούμενο κόσμο και σε διαρκώς τροποποιούμενες καταστάσεις. Ε, μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο συντονισμός, ενώ τώρα ε, βλέπουμε ότι ε, όλα διασυνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει μια κεντρική διασύνδεση με την Ατζέντα 2020, δηλαδή με αυτό που, προς το οποίο στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Και βεβαίω πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε ε, να στεφτούν από επιτυχία όλα αυτά τα βήματα. Ε, δηλαδή αποφασίζουμε πρώτα αν εφαρμόσουμε το πλαίσιο και αν το εφαρμόσουμε τότε συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για συνοχή, για συνεκτική μάλλον διαχείριση, για καλή διαχείριση, καλή διακυβέρνηση κτλ. Is key. over ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Γερουσίας είπε μερικά πολύ σημαντικά πράγματα. Όταν μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας για τους νέους, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει νέα πνοή ε, σε κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε προτείνει εμείς και στο παρελθόν. Και μία υποσημείωση. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ψήφισε ε, ε, ψήφισε μία έκθεση για την σύγκληση πολιτικών όσον αφορά δηλαδή το Ταμείο Συνοχής, Ταμείο ε, Γειτονίας αλλά εμείς διαπιστώνουμε ότι όσα σχετίζονται με τα εξωτερικά σύνορα δεν λειτουργεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να το πω. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Ε, και τα χρήματα τελικά επιστρέφουν στο ταμείο. Ε, γίνονται μεγάλοι προγραμματισμοί, ακούγονται πολλά πράγματα ε, κάνουμε ένα σωρό πράγματα για την Ουκρανία, για το Κίεβο, αλλά τελικά δεν ολοκληρώνονται. πολλά πράγματα λοιπόν ακόμα μπορούν να γίνουν και σίγουρα να μπει μια τάξη σε όλα αυτά. Λοιπόν, ε, μία πρώτη απάντηση σε αυτόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ε, επικοδομητικές ε, παρεμβάσεις που βέβαια άσκησαν και κάποια κριτική και αυτό το θεωρώ θετικό γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της ε, διαδικασίας και δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Θα έχουμε αρκετό καιρό να φωτίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σε ορισμένες ε, παρεμβάσεις διαπίστωσα ορισμένες ε, παρανοήσεις που ίσως σχετίζονται με το ότι οι αντιδράσεις ε, τελικά οι παρεμβάσει μάλλον των συναδέλφων αναφέρονται σε κάποια σχέδια προτάσεων που δεν έχουν προσλάβει ακόμα την οριστική τους μορφή. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα συχνά όταν ε, δουλεύουμε πάνω σε χαρτιά που δεν έχουν, όπως είπα, προσλάβει μια τελική μορφή. Αλλά είναι σχεδιάσματα. Ε, για παράδειγμα, ο φόρος προς θέμενες αξίας, το θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί οριστικά ερώτηση που τέθηκε από τον Ούγγρο εκπρόσωπο. Ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο εκπίπτει, θα εκπίπτει όχι. Ε, νομίζω ότι εδώ διαμορφώνουμε μια εσωτερική ευελιξία και αυτό είναι έκφραση των ε, διαφόρων πολιτισμών που εκπροσωπούνται εδώ και των διαφορετικών συνηθιών. Εδώ και μήνες έχω πει ότι θα λάβω χώρα στη Γαλλία σε μια περιφερειακή διάσκεψη και θα παρουσιάσω τις ε, ε απόψεις μου. Ε, τη θέση μου εδώ θα την ε, καλύψει ο Πέτε Μάρκοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους ε, συντάκτες του κανονισμού. και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο επιτελείο μου αλλά και στην υπηρεσία γιατί ε, εδώ πρόκειται βεβαίω για ένα τομέα της πολιτικής που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ε, συναδέλφους. Και ε, ήταν μια τεράστια πρόκληση να προσπαθούσουμε να βρούμε μια ισορροπία εν σχέση με τα, τις ανάγκες του προπολογισμού, σε συνάρτηση της ανάγκης του προπολογισμού. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, μπορείτε να βρείτε τις, ε, την τελευταία εκδοχή αυτών των κειμένων. Και παρακαλώ να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί θα ήθελα να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε πλήρως στη διάθεσή σας για, την, για οποιαδήποτε συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Και θα ήθελα να κάνω και μια άλλη παρατήρηση σε σχέση με μια ερώτηση η οποία τέθηκε εδώ το θέμα της μακροοικονομικής αρεσιμότητας που επανέρχεται σε πάρα πολλές συζητήσεις. Ε, θα ήθελα πραγματικά να σεβαστείτε το γεγονό ότι εντός της Επιτροπής ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα και δεύτερον ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών έχουν εξελιχθεί και τα, όλα αυτά τα θέματα και ε, πιστεύω ότι υποβάλαμε μία πρόταση ε, που είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά οφείλεται αυτό να γίνεται στη φύση της πολιτικής της συνοχής που είναι σύνθετη. Εάν διαβάσετε αυτή την πρόταση θα δείτε ότι πραγματικά αναφέρουμε την αιρεσιμότητα ως ίστατη προσφυγή εάν δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα άλλα μέτρα. Και αν πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας, μπορώ να κατευνάσω ανησυχίες των Έλλων συναδέλφων. Ε, στην παρούσα κατάσταση δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μακροαιρεσιμότητα. Γιατί όταν μια συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένη χώρα έχει ε, τεράστια οικονομικά, εκτοχιάζεται, αν θέλετε οικονομικά, υπάρχουν όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται με το Συμβούλιο και υπάρχουν πολύ εστιασμένες προτάσεις εν σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Και αν ε, μια χώρα μέλη ανταποκρίνεται σε αυτές τις προτάσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προστρέξει κανείς αυτούς τους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν αυτό το Sixth Pack, την ε, δέσμη των έξι μέτρων και ιδιαίτερως για τα μέλη της Ευρωζώνης ε, θεσπίζεται ένας μηχανισμός επιβολής ε, κυρώσεων. Εδώ έχουμε 17 χώρες μέλη στην Ευρωζώνη. Ελπίζω ότι θα είναι περισσότερα μελλοντικά και δεν θα πρέπει να έχουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το διαχωρισμό και νομίζω ότι θα ήταν πιο δίκαιο να πούμε ότι χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό ο οποίος να ισχύει και για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης αλλά όπως σας είπα ως ίστατη δυνατότητα προσφυγής, ultima ratio. Ε, και όσοι είναι παλιές καραβάνες εδώ ε, θα ξέρουν ότι από τότε που έχουμε ταμείο συνοχής εδώ υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση και μέχρι στιγμής για εύλογους ε, λόγους δεν έχει γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Λοιπόν, όπως σας είπα θα πρέπει να φύγω, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Παρακαλώ τον κύριο Βέσκοβετς να έρθει εδώ στη θέση μου. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε επικοδομητικές λύσεις. Και θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω την πολωνική κυβέρνηση, η οποία δείχνει μια ιδιαίτερη δέσμευση και ζήλο. Βεβαίως έχει και ήδη όφελος, αλλά αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω. Ο Πίτερ Μπέρκοβιτς συντόνισε όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Κομισιόν όσον αφορά την μελλοντική πολιτική συνοχή, σε όλο το κανονιστικό πλαίσιο. Οπότε, να ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές. Ο Δόκτωρ Χέλμουτ Μαρκόφ από τη Bundesrat, τη γερμανική Bundesrat. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής ιδιαίτερος όσον αφορά τις περιοχές τη πρώην Ανατολική Γερμανίας είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Γιατί στη διαδικασία μετασχηματισμού από την επανένωση το 1991 τα ταμεία, όλα τα ταμεία διαδραμάτισαν ένα τεράστιο ρόλο στην θετική υποστήριξη αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού. Και δεύτερον, τώρα ε, κατά πάσα πιθανότητα όλα τα ανατολικά κρατήδια θα φύγουν από την ε, κατηγορία στόχος 1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια εξυγένση του προπολογισμού, αλλά θα πρέπει επίσης να ε, στηρίξουμε μέσω πολιτικής συνοχής τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και νομίζω ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να τερματίσει αυτό το ρόλο κλειδί, γιατί ακριβώς είναι, έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και δεν είναι εστιασμένη στις βραχυπρόθεσμες ε, διακυμάνσεις της ε, οικονομίας. Ε, όσον αφορά τώρα την απομείωση, βεβαίως έχουμε πλήρη κατανόηση ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις για το phasing out. Όσον αφορά όμως το ύψος της συγχρηματοδότησης, εδώ θα πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε χώρες εκείνες που δεν έχουν επαρκή οικονομικά μέσα και δεν μπορούν να ε, καλύψουν αυτό το ύψος της δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Ε, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να προορίζονται δεν θα πρέπει να πέσουν για τις μειονεκτήσεις ε, περιοχές ε, κάτω από το 75%. Γιατί αν υπάρξει μία μείωση κάτω από το 75% ε, υπάρχει ο κίνδυνος η συγχρηματοδότηση να είναι τόσο υψηλή που να μην είναι εφικτή κάτω από την πίεση της εξυγίανσης του προπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές σύγκλησης που θα φύγουν από το στόχο 1 και θα πάνε στην ενδιάμεση κατηγορία, πώς ε, τεκμηρώνεται αυτή η ταξινόμηση. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να σας το πει η Επιτροπή. Ε, όπως σας είπα θα πρέπει να παραμείνουμε στο 75%. Ε, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η σταθεροποίηση. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που εμπίπτουν στο phasing out ε, θα πρέπει να θεωρούνται να εμπίπτουν στην μεταβατική κατηγορία. Αυτό αφορά ορισμένες κατηγορίες στη Γερμανία όπως είναι η λειψία ε, και άλλες που είναι αυτή τη στιγμή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και αν δεν υποστηριχθούν τελικά δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους γιατί δεν είναι ε, ε, επαρκές, ε, γιατί τα ποστά ενεργής είναι πολύ υψηλά, οι εκβιομηχάνες δεν είναι τόσο υψηλή κλπ. κλπ. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω να σκεφτείτε όλα αυτά τα προβλήματα και πάλι. Και τώρα τρία λεπτά για τον κύριο Αλφόνση κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο του Επιτρόπου Χαν μας βρίσκει σύμφωνο σε αρκετά σημεία όσον αφορά τις προτεραιότητες, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές, την πολιτική τα περιβάλλοντα. Είναι ένα κείμενο το οποίο αντιπροσωπεύει και για ένα βήμα, με ένα βήμα προς τα εμπρός, προς μια νέα αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής. Διότι το θέμα για μας είναι η πολιτική συνοχή στο μέλλον να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην εδαφικότητα και να μην ασχολείται μόνο με κάποια χάσματα ή στερήσεις συγκεκριμένων περιοχών. Θέλουμε μια εφορική προσέγγιση, θέλουμε κάτι αποτελεσματικό, επίσης όρις για όλους. Στο πλαίσιο αυτή τη πρόταση, οι ενδιάμεσε περιφέρειες είναι ενδιάμεσε ω προ την χρηματοδότηση και ω προς τα όρια για μας πρέπει να είναι ενδιάμεσες και όσον αφορά την ευελιξία των προγραμμάτων. Κάτι άλλο το οποίο μας δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες είναι η σύνδεση μεταξύ των εξαιρετικά αεροκατοικημένων περιοχών και των ε, εξόχως απομάκρων περιοχών. Η πολιτική μας συμπεριλάμβανε τα νησιά και τις ορεινές περιοχές. Γιατί χάθηκαν τα νησιωτικές περιφέρειες και οι ορεινές περιοχές. Μειώνεται έτσι, φοβούμε, η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο, εδαφική συνεργασία, έχουμε το συν 30%, λιγότερο από ό,τι περιμέναμε, αλλά και πάλι είναι μια αύξηση. Πιστεύουμε ότι η εδαφική συνεργασία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρότερη πολιτική βούληση και είμαστε υπέρ της ε, θέσπισης της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Τέλος, η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και περιφερειών πρέπει να είναι στο κέντρο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φοβούμαι ότι ο μηχανισμός κυρώσεων αποτελεί μια αντίφαση με τους στόχους μας. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι για τι ιστερίσεις τι οποίε υποτίθεται ότι πρέπει να θεραπεύσουμε. Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση. Θα παρέλθω όμω αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. επόμενο ομιλητή είναι ο κ. Λίνο Τουλίο από την ε, Επιτροπή προπολογισμού της Θελικής Βουλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να δραχθώ τη ευκαιρία και να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο έτσι όπως μας τα μετέφερε ο Επίτροπος κ. Ε, Χάν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά που ε, συχνά λέει ο καθηγητής ε, ε, Πρόντι που υπήρξε και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής <clears throat> όταν λέει ότι ολόκληρη η Ευρώπη, στο σύνολό της δηλαδή, είναι η πιο μεγάλη αγορά, είναι, έχει το μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα, αλλά ότι ξέχωρα η κάθε μία χώρα που την απαρτίζουν δεν έχει αυτή τη δύναμη δύναμη. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν της αναγέννησης της Ευρώπης ε, στην Τοσκάνη και στην ε, Κίνα ε, ενώ στη Ρώμη είναι η Γένοβα, είναι ε, χώρες, είναι πόλεις ε, οι οποίες στην αναγέννηση λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Μετά έγινε η πρώτη ανακάλυψη του νέου κόσμου, η Αμερική και από τη στιγμή που η Ιταλία μέσα από αυτές τις τόσο δυναμικές πόλεις δεν κατάφερε να ενωθεί όπως έκαναν άλλες χώρες όπως η Ισπανία, όπως η το Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν έτσι μια εθνική ε, δομή δεν κατάφεραν, έμεινε πίσω η Ιταλία. Ε, και συνεχίζει ο κύριος Πρόντι λέγοντας ότι εάν παραμείνουμε χωρισμένοι δεν θα καταφέρουμε ε, παρά ο καθένας ε, να κάνει ό,τι μπορεί για να επιπλέψει το καράβι του ενώ εάν ενωθούμε όλοι θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε πάρα πολύ δυνατοί. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε αλλά το πλαίσιο μπορεί να είναι καλό και όπως είπε και ο Γερμανός όμω, όμως ε, βλέπουμε πολλούς διαβόλου κρυμμένου στις λεπτομέρειες. Στο γενικότερο ε, πλαίσιο, εάν, ε, εάν βγάλουμε τα 39 εκατομμύρια της Connecting Europe Facility, βλέπουμε ότι φτάνουν σε 337 και Λυπούμε γιατί θα ήθελα να έχει υπάρξει αύξηση και όχι μείωση. Πιστεύω ότι η μείωση των ε, κονδυλίων ε, είναι αυτή η λογική του επαναπατρισμού ε, κεφαλαίων, τα οποία ορισμένες χώρες ε, θεωρούν ε, ότι είναι κακό και που, εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές λαμβάνει υπόψη κάποιες εθνικές πολιτικές. Γιατί, όπως λέμε και στην Ιταλία, καμιά φορά όταν κάνουμε κακές σκέψεις αμαρτάνουμε δύο φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση λίγο πιο πολύ Ευρώπη από τη μια μεριά, λίγο λιγότερο Ευρώπη από την άλλη ε, δεν είναι μια καλή πολιτική. Ε, ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός αφορά περίπου το 0,96% ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Ένα άλλο στοιχείο είναι αυτές οι μεταβατικές περιφέρειες ε, με 39 δις. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνουμε ε, καλά ε, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί, ποιος είναι ο λόγος δημιουργίας αυτής της νέας κατηγορίας, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια περικοπή της τάξης του 25% από τους στόχους σύγκλησης. Φαίνεται ότι μιλάμε ε, για 72 εκατομμύρια πολίτες ε, που όμως το μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκεται σε 5 ε, χώρες μέλη και επομένως αυτό το 75% των μεταβατικών περιοχών αφορούν μονάχα πέντε χώρες και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απολύτως αποδεκτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτά που λέω, ερωτήματα υποβάλλω, απλώς έχω την εντύπωση ότι ε, δίνονται περισσότερα, περισσότερα κονδύλια σε προθυμένες ε, χώρες ε, έτσι ώστε ακριβώς να επιστραφούν κεφάλαια τα οποία έχουν δοθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, βλέπω όμως, ε, ε, εκτός και αν κάνω λάθος, αλλά αναγυγνώσκοντας έτσι το, τη νέα δέσμη, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια εγγενής διαστροφή, γιατί εδώ δεν έχουμε ανακατενημητική πολιτική των πόρων μεταξύ των περιφερειών, αλλά μια πολιτική η οποία θέλει, προσπαθεί να αναπτύξει την εσωτερική αλληλεγγύη της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία θέλει ε, ο πρόεδρος Μπαρόζο δεν θα είναι δυνατόν να επιτύχουμε μια συνολικά ανταγωνιστικότερη οικονομία εάν δεν υπάρξει εσωτερική συνοχή. Ολοκληρώνω ε, αναφερόμενος ε, εις την μακροοικονομική ερεσιμότητα. θα είναι πραγματικά μία ultima ratio, όπως μας είπε ο Επίτροπος, αλλά πιστεύω ότι τέτοιου είδους διαφορετική προσέγγιση ενδεχομένως θα έχει κακό ε, αποτέλεσμα, θα ε, ζημιώσει τελικά ε, την, την πολιτική συνοχή γιατί είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλές οι χώρες και αυτό το είδαμε τώρα τελευταία, είναι πολλές οι χώρες οι οποίες αναγκάζονται να κάνουν κινήσεις διορθωτικές οι οποίες τελικά ζημιώνουν την πολιτική ανάπτυξη και όλες αυτές οι πολύ ωραίες συζητήσεις και τα πολύ ωραία λόγια ε, για ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, συνοχή κτλ. παραμένουν τελικά ωραία λόγια. Ε, η σωστή διακυβέρνηση που είναι ε, εκ των ουκάνευ προϋπόθεση για την συνοχή και την ανάπτυξη πραγματικά δεν εφαρμόζεται εδώ. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ συμπαθητικό όλα αυτά που λέω αλλά εν πάση περιπτώσει ε, η διασύνδεση με τη στρατηγική 2020 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως μπορεί ε, να συζητηθεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτή η διασύνδεση στις πλάτες, στο βάρος της πολιτικής ε, συνοχής. Βεβαίως πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν στο κεφάλαιο της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς ε, ε, γίνονται όλες αυτές οι αναφορές. Επίσης τα κριτήρια αναφοράς, οι δείκτες αναφοράς είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό που όμως μας αφήνουν λίγο προβληματισμένους. Οπωσδήποτε θα γίνουν, περιμένουμε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός και ελπίζουμε ότι με το νέο ε, κείμενο τουλάχιστον δεν θα επισοδρομήσουμε και δεν θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Σαγκουράκης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τη στιγμή που μιλάμε, που συζητάμε τα ζητήματα της ε, πολιτικής συνοχής, φαίνεται ότι η απόφαση της Ευρωζώνης του Ιουλίου για κούρεμα 21% του χρέους πάει ήδη για αναθεώρηση με ποσοστό κουρέματος έως και 50%. Τα λέω αυτά κυρία Πρόεδρε γιατί τα διέξοδα διαχείρισης της βαθιάς συγχρονισμένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καπιταλιστικής κρίσης όπως φαίνεται είναι αξεπέραστα. Ταυτόχρονα εντείνονται οι ανταγωνισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επιμερισμό της ζημιάς. Έτσι όλη η προπαγάνδα περί κρίσης χρέους και το αν αντιμετωπιστεί θα έρθει ανάπτυξη που θα ωφελήσει τους εργαζόμενους είναι κατά τη γνώμη μας κάλπικη. Τρόικα και ελληνική κυβέρνηση και κυβέρνηση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρεοκοπούν τους εργαζόμενους στην Ελλάδα με την καλπάζουσα ανεργία, τη δραστική μείωση μισθών, τη φορολιστία, τις περικοπές συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μία από τι αιτίε τη βαθιά κρίση στην Ελλάδα ήταν ασφαλώ και τα κοινοτικά προγράμματα που συνέβαλαν στην υπερσυσσόρευση κερδών για την πλουτοκρατία και στην γιγάντωση των ελλημάτων του ελληνικού κράτους λόγω των επιδοτήσεων στους βιομήχανους. Η πολιτική ε, συνοχή που συζητάμε σήμερα εξυπηρετεί την επιδίωξη των ευρωενωσιακών μονοπωλίων να συνδέσουν ακόμα πιο στενά την περιφερειακή πολιτική με την αντιλαϊκή στρατηγική Ευρώπη 2020, ώστε αυτή να υπηρετεί πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά την κερδοφορία τους. Έτσι, τα κονδύλια των 336 δις από το Ταμείο Συνοχής θα προσθεθούν στα ήδη 4,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραξαν οι τράπεζες στο όνομα της αντιμετώπισης της καπιταλιστικής κρίσης. Εγκαταλείποντας ακόμα και τις φραστικές δεσμεύσεις για την συνοχή των περιφερειών, επιλέξιμα θα είναι όλο και περισσότερο μόνο εκείνα τα προγράμματα που προωθούν ακόμα πιο αποφασιστικά την ενιαία αγορά και το σύμφωνο ε, Ευρωπλάς, δηλαδή εκείνες τις πολιτικές που οδήγησαν στη σημερινή καπιταλιστική κρίση. Επιδιώκεται η αδιανομή των πόρων που αφαιρούνται από τους λαούς μέσω από τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε υποδομές και έργα που εξυπηρετούν άμεσα ή έμεσα την ακόμα φθηνότερη εργατική δύναμη και νέες αγορές για την πράσινη τεχνολογία. Αυτό φαίνεται και από τις εξελίξεις στο ελληνικό ΕΣΠΑ, όπου η μείωση της εθνικής συνεισφοράς συνοδεύτηκε από την κατάργηση εκατοντάδων άλλων χρήσιμων για τη χώρα προγραμμάτων. Τέλος, επιλέξιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πρόκειται ποτέ να είναι έργα που ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες. Έργα για την αντισυσμική θωράκιση, την αντιπλημμυρική προστασία, τη λαϊκή κατοικία, την κατασκευή υποδομών για δωρεάν και αποκλειστικά δημόσια παιδεία, υγεία, πρόνοια, φτηνές και ασφαλείς συγκοινωνίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ. Πορτογαλία. Πέτρος, Πέτρος Άιβα. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Από την πλευρά μας πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Τρεις παρατηρήσεις όμως. Πρώτον, απλούστευση, κοινοί κανόνες, ανεξαρτήτως διαρθρωτικού ταμείου. Αυτό όντως σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συνοχή. Δεύτερον, για τις ε, περιφερειές μετάβασης, η κεντρική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον μηχανισμό, την εξέλιξη μάλλον του μηχανισμού phase in και phase out. Αλλά δεν θέλω αυτό να επιβαρύνει τις περιφερειές μας. Θα το δούμε αυτό. Τρίτον, επιτρέψτε μου να επανέλθω στην ομαδοποιημένη διαχείριση των προγραμμάτων. Με ενδιαφέρουν εδώ τα πολυταμιακά προγράμματα. Εκεί χρειαζόμαστε μια ενιαία διαχείριση, ανεξαρτήτως ταμείου. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση. Αλλά και τα άλλα που είπα πιστεύω ότι είναι σημαντικές προκλήσεις και θα περιμένω κάποιες απαντήσεις. Επίσης, όσον αφορά τη νέα πρωτοβουλία Connecting Europe, συμφωνώ με την γενική κατεύθυνση αν και θα κοστίσει αρκετά. Απορροφάμε δηλαδή έτσι ένα κομμάτι του Ταμείου Συνοχής. Τουλάχιστον να σας διασφαλίσουμε την άλλη πλευρά ότι η ενιαία διαχείριση θα αρισταθμίσει αυτή την απώλεια. Δεύτερον, πρέπει η πολιτική συνοχής να συναρθρωθεί με την πολιτική 2020. Όμως, δεν θέλω να βάλουμε την εδαφική συνοχή σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Στην στρατηγική 2020 δεν υπάρχει σαφής σύνδεση με την εδαφική συνοχή και δυστυχώς υπάρχουν δύο διαφορετικές λογικές ως προς αυτό. Με άλλα λόγια, δεν θέλω η εδαφική συνοχή να είναι παραπέδι της στρατηγικής για το 2020. Να είναι ο φτώχος συγγενής, αν θέλετε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, γνωρίζουμε όλοι ότι στην περασμένη προγραμματική περίοδο χρειαστήκαμε δύο ολόκληρα χρόνια. 2007-2008 οι μηχανισμοί δεν ήταν έτοιμοι, οπότε απευθύνω έκκληση εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου να βιαστούμε. Ο χρόνος πιέζει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Ευχαριστώ πολύ. Στους συναδέλφους που φεύγουν, ε, μην ξεχνάτε ότι θα πιούμε ένα ποτήρι μαζί αμέσως μετά, στις 6.30. Ε, Ο πρώτος ομιλητής δεν είναι εδώ. Έρικα Ρίξον από Σουηδία, από την Σουηδική Βουλή. Η πολιτική συνοχής ήταν και θα είναι χρήσιμη. Αλλά ας μην ξεχνούμε και την άλλη αρχή της επικουρικότητας. Το λέω αυτό διότι καταρχήν τα κείμενα δεν έχουν μεταφραστεί, άρα τι να πω. Είναι όμως ενδιαφέρον να ακούω τουλάχιστον τους άλλους ομιλητές. Παρά τη δυσκολία συμμετοχής σε αυτήν την συζήτηση. Αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων, ναι, φυσικά, είναι πολύ χρήσιμο. Και είναι σημαντικό για την πολιτική συνοχής, όπως και για την γεωρική πολιτική. Πρέπει όμως να συνδέσουμε όλα αυτά τα συστήματα μεταξύ τους, γιατί σε κάποιες περιοχές τα πράγματα λειτουργούν ικανοποιητικά, όχι όμως παντού. Χρειαζόμαστε επίσης καινοτομία στην περιφέρεια. και ξέρουμε ότι προς τούτο χρειάζεται βοήθεια από το κέντρο. Αυτήν την πολιτική θέλουμε να προωθήσουμε. Η έλλειψη κεφαλαίων βεβαίως είναι πρόβλημα. Οι τελείς συνάδελφοι το έθιξαν το ζήτημα αυτό. Ξέρετε, το αισθανόμαστε και εμείς, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες δεν στέκονται στο ύψος των ευθυνών τους. Δεν θέλουμε λοιπόν λόγω έλλειψης κονδυλίων να δοθεί μάχη μεταξύ των περιφερειών με σύνθημα θανατώσου η Η ζωή μου. Τώρα στον ε, τομέα της καινοτομίας ας αλληλοβοηθηθούμε. Ξέρετε, σε ορισμένες περιφέρειες υπάρχει τρομακτικός ανταγωνισμός. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα και γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα. Έχω μάλιστα μία ερώτηση και δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε. Αφορά το χρονοδιάγραμμα και δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις τέλη Οκτωβρίου, είναι σωστό αυτό, είναι ακριβές, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Διότι πρέπει καταρχήν να μεταφραστούν ένα σώρο έγγραφα και φυσικά μετά πρέπει να γίνει η συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια και ούτω καθεξής. Περιμένω λοιπόν μια απάντηση. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που είναι ο Επίτροπος εδώ. Αυτά προς το παρόν ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω, άρα Πορτογαλία και πάλι. Μαρία Ελένα Ανδρέα από την Πορτογαλική Βουλή. Κυρία Πρόεδρε, θα συγχαρώ και εγώ την κυρία Χιούμπνερ για την διοργάνωση αυτής της σύσκεψης αρκετά νωρίς πριν από τις τελικές αποφάσεις. Από ό,τι άκουσα, υπάρχουν τρεις θεματικοί τομείς, τρεις θεματικές ενότητες που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια της συζήτησης. Πρώτη θεματική ενότητα. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στη θετική στάθμιση των διευθυντικών πολιτικών ως τώρα. Ήταν η μόνη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τώρα είμαστε αντιμέτωποι με τόσες αβεβαιότητες στο μέλλον. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πολίτες διερωτώνται τι προστιθέμενη αξία έχει η Ευρώπη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η πολιτική συνοχή να είναι ορατή, αλλά κυρίως, επί της ουσίας, να κάνει τη διαφορά σε σύγκριση με το παλιό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Και το νέο πρέπει να είναι υπέρ του κοινωνικού μοντέλου ανάπτυξη για τι χώρε μα και τι περιφέρειε. Πρέπει, όπω ε, προείπα, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό είναι θεμελιώδε ζήτημα. Ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, εν προκειμένου, θα είναι επίση πολύ σημαντικό. Α αφήσουμε κατά μέρο του εθνικού εγωισμού, α προσεγγίσουμε τι πολιτικέ μα αν θέλουμε να προχωρήσει η Ευρώπη. Τώρα για άλλα ζητήματα υπάρχει λιγότερη συνένεση. Το πρώτο είναι τι προσδοκούμε από την κοινωνική, οικονομική και δαφική συνοχή. Δεν βλέπουμε όλοι μας το θέμα με τον ίδιο τρόπο. Παρά στο βέβαιο είναι ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χαρακτηρίζεται πλέον από σαφέστερα καθορισμένους στόχους που συνάδουν με τη στρατηγική 2020. Και τούτο παρά την μεγαλύτερη ευελιξία που θα έχουμε από εδώ και πέρα προς τις μεθόδους. Η αλήθεια είναι ότι αυτόν τον καιρό εξευρωπαίζουμε, αν θέλετε, κάποιες εθνικές πολιτικές. Αυτό είναι καλό. Έτσι θα είμαστε πιο κοντά στους στόχους μας. Με αυτήν την οπτική εν γέννη συμφωνώ. Όμως χρειάζεται και εδώ προσοχή. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της παραδοσιακής αλληλεγγύης των διαρθρωτικών ταμείων και των νέων προτεραιοτήτων και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν κράτη-μέλη και περιφέρειες. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι η Ευρώπη το 2014 όταν θα αρχίσει να ισχύει το νέο πλαίσιο. Ίσως έως τότε να έχουν προκύψει νέες προτεραιότητες οι οποίες ε, θα προσθεθούν στα σημερινά προβλήματα. Πέραν αυτών, συμφωνώ ότι έχουμε δύο άλλα ουσιώδη ζητήματα που πρέπει να μας προβληματίσουν και σε εθνικό επίπεδο. Το πρώτο είναι οι ερεσιμότητες όπως λέγονται, τα conditionalities, ως προς την χρήση των ταμείων. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην χρήση των πόρων και επίσης υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά το αποθεματικό αποτελεσματικότητας. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να θέτουμε σε δυσμενέστερη μοίρα με δύο διαφορετικούς τρόπους τις ίδιες περιοχές. Επειδή ενδεχομένω κάτι δεν πήγε καλά στην εταιρική σχέση μεταξύ κράτου μέλους και κομισιών. Αλλά ξέρετε, εκεί μπορούν πολλά πράγματα να μην πάνε καλά. Γι' αυτό πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και να βρούμε ένα κοινό τόπο. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχω ορισμένε αμφιβολίες όσον αφορά τη μείωση των πόρων που διατίθεται στις πιο φτωχές περιοχές μέσω της δημιουργίας της ενδιάμεσης κατηγορίας. Δεν λέω, τα κονδύλια πρέπει να πάνε παντού, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα ευρύτερα και να δούμε εν τέλει πώς θα βγούμε από την κρίση, γιατί αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αντιμετωπίζοντας βεβαίως και τους ε, κινδύνους που αντιμετωπίζουν πιο φτωχές περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, Σαν Κελή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η πολιτική συνοχή, δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν πολύ επιτυχή. Πολλέ περιφέρειε επωφελήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη η αναθεωρησή της λόγω της κρίσης. Η πρώτη παρατήρηση είναι, αν δω τα εθνικά κοινοβούλια που εκπροσωπούνται, λέει, 13. Πού είναι τα άλλα 14, δεν τους προσκαλέσατε κυρία Πρόεδρε ή δεν ήρθαν απλώς. Δεύτερον, άκουσα πολλά για την ενδιάμεση κατηγορία των περιφερειών. Κάποιοι αντιδρούν. Πιστεύω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα στην Επιτροπή Επιτροπή μας, στο Κοινοβουλίο γέννη. Αυτοί που είναι υπέρ, δεν νομίζω ότι μπορούν να κατηγορηθούν ότι το κάνω από εγωισμό για να εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα. Ούτε είναι αλήθεια ότι θέτουμε σε δυσμένες θερμίδια τις πολύ φτωχές περιοχές μόνο και μόνο επειδή για κάποια πεπερασμένη περίοδο οι περιοχές μεταξύ 75% και 90% του κινητικού μεσοόρου λαμβάνουν μια ειδική ευνοϊκή μεταχείριση. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα, άξια συζήτησης. Τέλος, επειδή ακούσαμε και την ευελιξία για τις περιφέρειες, η κατηγοριοποίηση μου φαίνεται λίγο αυθαίρετη και αναχρονιστική σε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν μάλλον ευελιξία και στην κατηγοριοποίηση των περιφερειών. Τα όρια λοιπόν να επανασχεδιαστούν αν θέλετε. Τα όρια των ίδιων των περιφερειών σε ορισμένε περιπτώσει δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Σε ορισμένε περιπτώσει θα έπρεπε ενδεχομένω να επανασχεδιαστούν. Χιούμπνερ, Κύπρος, ο κύριο Χατζηγιάννης. Παρακαλώ. Επιτρέψατε να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να δεσμευθούν οι, βουλευτικοί όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, σήμερα τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονομεύει την ε, απτή πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής η κρίση έχει υπογραμμίσει τη δυνατότητα οι ανισότητες να αυξηθούν. Και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη μιας εναρμόνισης της ανάπτυξης της Ευρώπης η σημασία της πολιτικής συνοχής είναι όλο και πιο προφανής, όχι μόνο για να μετρεστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, αλλά επίσης σαν ένα εργαλείο οικονομικής αναζωογόνησης. Οι χώρες μέλη τώρα αντιμετωπίζουν πολλές ε, δυσχέρειες, πολλά προβλήματα και έχουν βεβαίως λογικές προσδοκίες από την πολιτική συνοχής. Μεταξύ αυτών και δική μου η χώρα, η Κύπρος η Κύπρος έχει προσφύγει στο Ταμείο Αλληλεγγύης μετά από μια έκρηξη, μια ναυτική βάση που ζημίωσε πάρα πολύ τον, το σταθμό ηλεκτρικής, ε, τη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδότησης της χώρας. Ένας ε, ε, πολλές χώρες μέλη πιέζουν το Ταμείο Συνοχής γιατί ε, και επίσης τα, η υπερχρέωση πολλών ε, χωρών ε, δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τα κριτήρια της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης στα οποία βασίζονται τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Υπό την έννοια αυτή, η ενθάρρυνση του του ιδιωτικού κεφαλαίου είναι προϋπόθεση για την είναι σημαντική όσον αφορά την ε, πολιτική συνοχή. Μέσω της ε, Ευρώπης 2020 ε, μπορούν να επιτευθούν οι σκοποί μιας βιώσιμης ανάπτυξης, αλλιώς θα παραμείνουν κενό γράμμα. Η ισχυρότερη διασύνδεση πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και η στίεση στα περιεχόμενα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής και καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί αρκετή προσοχή ούτω ώστε να μην υπονομευθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών και επίσης οι, οι διαχειριστικές δυνατότητες κάθε χώρας μέλους. Ε, όλα αυτά διαφωνούν την... Ε, ε, ε, όλα αυτά πρέπει να επίσης με την αρχή της επικουρικότητας και της αξίας που προβάλλει το κάθε εθνικό κοινοβούλιο. Ο χαρακτήρας της πολιτικής συνοχής δεν θα πρέπει να περιορίζεται υπέρ μιας τομεακής προσέγγισης γιατί η πολιτική αυτή είναι διατομεακή και αυτό είναι ένα από τα βασικά της κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερο σημαντικός και δεν θα πρέπει να εξαντλείται στον έλεγχο της επικουρικότητας στην νομοθετική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι στόχοι της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, επιτυγχάνονται και υπάρχει μια αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πίτερ Μπέρκοβιτς από την Επιτροπή. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια ε, τα, και τις ερωτήσεις που άκουσα. Βεβαίως ε, δεν θα μπορέσω, δεν έχω το χρόνο, γιατί άλλωστε έχετε και μια δεξίωση, δεν έχω το χρόνο να απαντήσω. Ε, εν πάση περιπτώσει, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Το πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα να αντιμετωπίσω είναι το θέμα της εμπλοκής των περιφερειών. Θα ήθελα να είμαι κατά αυτή την έννοια πάρα πολύ σαφής. Η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική η οποία στηρίζεται σε διακυβέρνηση πολυεπίπεδη οργανώνεται από τα κράτη-μέλη και θα ε, συνεχίσει να είναι έτσι. Βεβαίως θα υπάρξει μηχανισμός ε, συντονισμού που όμως δεν θα αντικαταστήσει τα μέχρι τώρα ισχύοντα προτείνουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς ε, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή και θα ε, εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη και τους εταίρους ε, στην δημιουργία εταιρικών σχέσεων. Και νομίζω λοιπόν ότι ε, είναι ε, ε, σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Δεμπέργκ, να δούμε το σύστημα των ελέγχων. Εδώ θα πρέπει να εξισορροπηθούν σωστά τα πράγματα. Από τη μία πλευρά έχουμε το κόστος της τοπικής και εθνικής διαχείρισης και από την άλλη πλευρά έχουμε την ε, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στις αρχές επί του προϋπολογισμού ε, που θα πρέπει να καταδείξουν ότι γίνεται σωστά ε, η διαχείριση των πόρων. Uh, θα θέλαμε να προτείνουμε έναν μεγάλο ρυθμό απλουστεύσεων που πιστεύουμε ότι θα μειώσει το συνολικό κόστος, αλλά θα μειώσει οπωσδήποτε και τις περιοχές, αλλά και το ποσοστό σφάλματος. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ένα σωστό σύστημα ε, που ε, θα αφορά αυτό που παλιά λέγαμε συμμόρφωση και τώρα ονομάζομαι πιστοποίηση. Ε, πιστεύουμε επίσης ότι στο ίδιο το σύστημα ελέγχων ε, ο εξωτερικός οικονομικός έλεγχος θα πρέπει να ε, μπορεί να προσαρμόζεται κατά περίπτωση. Όσον αφορά το ζήτημα της ανάμειξης των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, κάποιοι μεταξύ ημών αναφερθήκατε στο urban Ε, από την άλλη πλευρά εμείς ε, προτείνουμε μια προσέγγιση της ε, τοπικής ανάπτυξης που συνάδει περισσότερο με την αρχή. Δυστυχώς υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα μέσα στην αίθουσα, δημιουργούν μεγάλες παρεμβολές. Θα θέλαμε ε, να δώσουμε μια νέα κινητροδότηση αν είναι δυνατόν. Ε, γιατί θέλουμε λοιπόν μια νέα, ε, μια νέα μορφή μεταβατικών περιφερειών. Πολύ απλό γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το, το σύστημα που προτείνουμε είναι πιο δίκαιο από το υφιστάμενο, το ισχύον σύστημα. Ε, στο ισχύον σύστημα, ε, εάν έχετε μία περιφέρεια η οποία είναι ε, του 250% του ΑΕΠ, τότε θα πάρει τα ίδια χρήματα με μια περιοχή της τάξης του 76% ΑΕΠ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δίνοντας, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία 75-90, τότε ε, πραγματικά δημιουργούμε ένα ε, δικαιότερο σύστημα αλλά επίσης ε, και ένα δίχτυ ασφαλείας για τις περιφέρειες εκτός σύγκλησης. Όμως να καταστήσω σαφές ότι δεν προβλέπουμε μονάχα ένα δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά την χρηματοδότηση αλλά και όσον αφορά τη συγκέντρωση πόρων. Να πω δύο λόγια σχετικά ε, με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ε, στον κανονισμό, εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το υφιστάμενο σύστημα. Στρέφομαι στο ζήτημα των οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ετέθησαν ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την εγκυοδοσία τους, τα μία κτλ εμείς ε, προτείνουμε διάφορα εργαλεία τα οποία πιστεύουμε ότι θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, να προστρέξουν ε, σε δυνατότητες οι οποίες υφίστανται ήδη και επομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για πολλές δραστηριότητες τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα. Ε, προγράμματα πολλαπλής ε, χρηματοδότησης ή χρηματοδότηση από πολλά ε, ταμεία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, όχι όμως σαν υποχρέωση. Δηλαδή, αν κάποια χώρα θέλει να συνεχίσει με προγράμματα ενός χρηματοδότησης ενός ταμείου, μπορεί να το κάνει. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της Ευρώπης 2020, Αυτό που θα θέλαμε στο μέλλον είναι μεγαλύτερη εστίαση στους στόχους της Ευρώπης 2020. Τι σημαίνει αυτό. Το καθιστούμε σαφές στον κανονισμό. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη δουλειές, θέσεις εργασίας ε, και κάποιους άλλους στόχους που συνδέονται με το 2020. Αλλά το πώς, ο τρόπος επίτευξης των στόχων αυτών αφήνεται ανοιχτός. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν πολλαπλές λύσεις ευθυγράμμισης με τους, ε, με τους στόχους 2020 να βρεθούν λοιπόν λύσεις που θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες και θα είναι σωστές για τις δικές σας περιφέρειες, για τις δικές σας ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε και στις διαπραγματεύσεις και στα προγράμματα να έχουμε διαρκείς επαφές μαζί σας. Αυτή είναι άλλωστε η προστιθέμενη αξία αυτού του προγράμματος συνοχής. Είναι απολύτως θεμελιώδους σημασίας. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της χωρίς τοπικές και περιφερειακές λύσεις και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση στο μέλλον για τα ζητήματα αυτά. το αποθεματικό αποδοτικότητας ή απόδοσης performance reserve αυτό ε, το προβλέπουμε σε εθνικό επίπεδο όταν υπάρχει ένα αποθεματικό για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις που έχουν επιτευχθεί ε, οι στόχοι και εμείς ε, λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο τα προγράμματα τα οποία λειτουργούν καλύτερα κάποια στιγμή να τύχουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση Πάντως μπορούν να βελτιωθούν οι αποδόσεις. Όσον αφορά το θέμα της συγκέντρωσης, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συγκέντρωση αλλά η συγκέντρωση αυτή οπωσδήποτε θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ε, χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης ε, για τις περιφέρειες σύγκλησης. Λέμε επίσης ότι ε, οι περιφέρειες οι οποίες τώρα βγαίνουν από την, από την σύγκληση που είναι λιγότερο από 70% εκεί θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή του ποσοστού συγκέντρωσης απόσυρση των ε, ε, ορίων τα όρια τα οποία δίνει, ε, ορίζει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ΝΑΤΣ κτλ. Βεβαίω, αν κάπου υπάρχει παραλογισμός, οπωσδήποτε τα κρατημέλη μπορούν να τροποποιήσουν κάτι. Τέλος, τελευταίο σημείο. Ε, το τελευταίο μου σημείο λοιπόν αφορά την εγκάρσια προσέγγιση. Ε, πιστεύω ότι έχουμε δώσει την βάση για μια ε, στενότερη σχέση ανάμεσα στο Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΚΤ και τα τα πολυταμιακά προγράμματα. Μία νέα προσέγγιση, κοινοτική, ενωσιακή προσέγγιση που θα δώσει την δυνατότητα να εφαρμοστεί ε, ένα σύνολο κανόνων, ε, όχι μονάχα στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στην, ε, στους θαλάσσιους πόρους, στη γεωργία κτλ. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Να σας πω ότι αυτή είναι μια νέα εμπειρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που εμείς προτείνουμε προτείνουμε, κάνουμε πρόταση ε, για τη συνοχή υπό την ε, τροποποιημένη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει ένα πρώτο έναυσμα συζήτησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια που ευελπιστούμε ότι η συζήτηση αυτή θα είναι μακρά και καρποφόρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ ως αρμόδιος του Bundesrat. Ε, μου δίνει ως του Bundesrat. Θα ήθελα να επισέλθω δύο σημεία της συζήτησης. Η, Γερμανική Βουλή τις επόμενες εβδομάδες θα εκδώσει μια περιεκτική γνωμοδότηση για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτή η γνωμοδότηση θα μεταφραστεί και θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ρέγγι. Ε, τα κρατήδια συμφωνούν με την γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο ότι οι προτάσεις ε, ε, είναι επαρκής όσον αφορά την ανάγκη συγκέντρωσης. Ε, υπήρξαν οι συνεδριάσεις της ΚΟΖΑΚ πριν από μερικές εβδομάδες και ορισμένοι εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων έθεσαν αυτό το θέμα να της συγκέντρωσης. Αλλά 72% των κονδυλίων πρέπει να προορίζονται για τις πιο αδύναμες ε, περιοχές. Και είναι 27 περιφέρειες ε, οι οποίες θα εγκαταλείψουν το στόχο σύγκλησης στην προσεχή περίοδο. Και αν λάβουμε όλα αυτά υπόψη μπορούμε να πούμε ότι οι προτάσεις της ε, ε, επιτροπής πράγματι εστιάζουν στις πιο αδύναμες περιοχές, κάτι που επιθυμούμε και εμείς. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει η πολιτική της συνοχής μελλοντικά να ε, ε, παραμένει ανοιχτή προς όλες τις ε, περιφέρειες και αυτό συνδυαθήνει με την Ατζέντα 2020 γιατί η συνοχή πολιτικής μπορεί να κάνει πολλά για την ελοπίση στρατηγική 2020 αλλά δεν πρέπει να περιοριστεί στις πιο αδύναμες περιφέρειες αλλά θα πρέπει όπως σας είπα να προσφέρει σε όλες τις περιφέρειες και όλες οι περιφέρειες διαβαθμισμένα πρέπει να συμμετέχουν στα διευθυντικά ταμεία. Τέλος, όσον αφορά, τελευταίο σημείο όσον αφορά τις μεταβατικές ε, περιφέρειες. Έχουμε το πρόβλημα της μετάβασης, δηλαδή οι σημερινές περιφέρειες σύγκλησης που λόγω μιας θετικής ε, εξέλιξης βρίσκονται πάνω από το κατόφλι του 75%. Δηλαδή 16 περιφέρειες σύγκλησης, 11 περιοχές phasing out που αυτή τη στιγμή παίρνουν χρήματα από το Ταμείο Ε, και έχω την άποψη και το ίδιο και η γερμανική κυβέρνηση ότι αυτές οι περιφέρειες θα πρέπει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να παίρνουν κάποιες μεταβατικές ενισχύσει. Τα άλλα στα οποία ασκήθηκε κριτική εδώ είναι ο νέος στόχος να περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες ε, που βρίσκονται μεταξύ του 75% και 90%. Αυτό είναι που δεν θέλουν οι Γερμανοί, γιατί θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό ορίζεται ένας νέος στόχος, όπου τελικά δεν βλέπουμε που βρίσκεται ακριβώς η διαφοροποίηση στο σημερινό στόχο της ανταγωνιστικότητας. Ε, πού γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Γι' αυτό λέμε μεταβατική ενίσχυση ναι, ε, δύο τρίτα των σημερινών ε, κονδυλίων, αλλά πραγματικά μια προσεκτική εξέταση του ενδιάμεσου στόχου, αυτού που βρίσκεται δηλαδή στο στο 75 και 90%. Φτάνουμε στο τέλος της συνεδριασής μας. Επιτρέψτε μου να σας καθυστερήσω δύο-τρία λεπτά για να σας πω ότι καταρχήν θα τα πούμε σε ένα χρόνο από σήμερα με την ίδια σύνδεση. Σύνθεση, με συγχωρείτε. Αυτό αποφασίσαμε θα ξαπούμε, Οκτώβριο του 12. Και ελπίζουμε ότι τότε θα είμαστε πολύ πιο κοντά στην απόφαση που αφορά το νέο κανονιστικό πλαίσιο και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ανάπτυξη θα έρθει από τις περιφέρειες, από τις πόλεις, την καινοτομία. Αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε. Θέλουμε να δούμε νέα επενδυτικά σχέδια να χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής από το, 2014. Το οποίο είναι αύριο, γι' αυτό και βιαζόμαστε. Η Κομισιόν, αλλά και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γραμματεία... Ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα σχόλια. Ήδη σύντομα θα έχω τα σχόλια σας και εκτυπωμένα. Λοιπόν, Ακούσαμε πολύ προσεκτικά να ξέρετε, αλλά όποιος θέλει να στείλει και κάτι άλλο γραπτός, είμαστε όλα αυτιά. Ούτως ή άλλως τώρα ξεκινάει αυτή η συνεργασία. Όπως είπα στην αρχή, έχετε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα για τον ελέγχο επικουρικότητα στα χέρια σας, αλλά δεν είναι το θέμα να φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι να συνεννοηθούμε, να δούμε τι μπορείτε να κάνετε εσεί, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί. Και υπάρχουν και επιτροπέ στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία ασχολούνται με διαπραγματεύσει, δημοσιονομικού χαρακτήρα ή σχετικά με άλλε πολιτικέ. Έχετε και εσεί τη δική σα δραστηριότητα. Προσβλέπουμε επίση την ε, συνεργασία σα με τι κυβερνήσει, γιατί κάποιε κυβερνήσει εισακούν και τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να επηρεάσετε τι δικέ σα κυβερνήσει ο καθένα στη χώρα του εξού σημαντικό για όλους μας. Επίσης, θα ήθελα να πω, όπως προείπα, ότι τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύουμε πολύ σκληρά εν ώψη αυτής της διαπραγμάτευσης, εμπιστοσύνη με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο, προτιμάζοντας ψηφίσματα, ψηφίζοντας την Ολομέλεια, ενημερώνοντας συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι σημαίνει η συνοχή και συνεργαζόμαστε και μια ειδική επιτροπή εργασία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Είμαστε στην Κομισιόν προημερών. Γίνονται πράγματα δηλαδή. Επίσης, ορίσαμε εισηγητέ για όλες τις ε, πολιτικές. Έχουμε εισηγητέ από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες, από το ΕΛΚ, ε, τον Λάμπερτ Φανιστερόι, τον Τσέλερ, ε, από τη Γερμανία την Πολωνία και την Ολλανδία, από τις σοσιαλιστές είναι λοιπόν, Μποστινάρο από τη Ρουμανία και η Μαρία Ριγκόγεν Πέρες από την Ισπανία και την Κωνσταντζα Κρέλ από τη Γερμανία και από τους φιλελευθέρους έχουμε την Έρικα Μάνερ από την Φινλανδία. Πάντως να ξέρετε ότι για κάθε εισηγητή υπάρχουν και σκιώδεις εισηγητές από άλλες πολιτικές ομάδες. Αν ε, αισθάνεστε πιο άνετα να μιλήσετε με τη δική σας πολιτική οικογένεια, μπορείτε να έρθετε σε επαφή είτε με εμά είτε με τους συγκεκριμένους συναδέλφους που ανήκουν στη δική σας πολιτική ομάδα. Όλη η πληροφορία αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, τόσο ή άλλως. Η η σύσκεψή μας είναι σε ένα μήνα από σήμερα, οπότε θα ανταλλάξουμε απόψεις και πάλι για το μέλλον του κανονιστικού πλαισίου. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό όμως. Υπολογίζουμε σε εσάς γιατί μαζί είμαι βεβαία ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι θα πορευτούμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Ο μόνος δρόμος είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος. Με αυτά θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε να πάρουμε ένα ποτήρι μαζί και κηρύσω το πέρας της συνδριάσεως. Μετά τους Πολωνούς σας υπενθυμίζω ότι έχουμε Δανική Προεδρία και μετά Κυπριακή Προεδρία. Οι Πολωνοί κάνουν πολύ καλή δουλειά. το ξέρετε αυτό για να μιλήσετε με τους ε, αριστείχους συναδέλφους από τα αντίστοιχα κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που ήρθατε. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε στον καλό δρόμο που χαράξαμε. Καλό σας βράδυ.